There is work still to do, but we are aiming to meet at least the level of ambition as set out by the group of personalities in its report that the future European Defence Research Programme will need a total budget. Θα χρειαστεί προϋπολογισμό 3,5 δισεκατομμυρίων τουλάχιστον για το, για το διάστημα 2021-2027 προκειμένου να είναι αξιόπιστη. Παρά το γεγονό ότι η έναρξη του επόμενου προγράμματος Κομισιόν ε, ε, θα ξεκινήσει σε πέντε χρόνια, ε, θα πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι ε, θα ε, επηρεάσει και τον οργανισμό μας αλλά και τις ικανότητες των κρατών μελών. Πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό στα ισχύοντα τα υπάρχοντα προγράμματα των κρατών μελών. Πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η οριστικοποίηση της... στρατηγική αυτή θα ανοίξει ε, μία σειρά από δυνατότητε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με βάση ε, τη δουλειά που έγινε για την ασφάλεια και την άμυνα, ο οργανισμός μας θα πρέπει να αναθεωρήσει την, ε, τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ανάπτυξη στρατιωτικού δυναμικού και στην ουσία και στην ε, μεθοδολογία. η CDP είναι ο φορέας αναφοράς για αυτή την ανάπτυξη. δίνει ουσιαστικές δυνατότητες και στο ΝΑΤΟ για τον αμυντικό σχεδιασμό, γιατί κάθε κράτος μέλος έχει ε, τις μοναδικές δικές του δυνάμει ε, σε συμφωνία με τον ΝΑΤΟ και θα πρέπει να συνεχίσει ε, αυτή την προσπάθεια. Εμείς ε, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη πολυεθνικού ε, στρατιωτικού δυναμικού γιατί τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επενδύουν περισσότερο και περισσότερο μαζί σε στρατιωτικό δυναμικό. Ε, θα πρέπει να κλείσουμε τα κενά που υπάρχουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο ανεφοδιασμο αερος αέρος-αέρος που είναι ε, βασική προπόθεση για την ε, προβολή αεροπορικής ισχύω και είναι σημαντικό για να υπάρχουν επιχειρήσεις στον αέρα ε, μάχες δηλαδή, ε, οι οποίες κρατάνε πολύ. Στο παρελθόν οι Ευρωπαίοι ε, βασίστηκαν συστηματικά σε αμερικανικέ αμερικανικές δυνάμεις, στρατιωτικά μιλάω. Αυτό επιβεβαιώθηκε το, το δίδαμε στο Κοσμοπέδιο το 1999 και επιβεβαιώθηκε στη Λιβύη το 2011. Στην επί... οργανισμό μου έχουμε τρεις στόχους. Να αυξήσουμε το δυναμικό ε, ανεφοδιασμού αέρος-αέρος, να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό ε, του ευρωπαϊκού ε, στόλου ε, τάνκερ και να βελτιστοποιήσουμε τα υπάρχοντα ε, στοιχεία που έχουμε, εργαλεία, οργανώσεις κτλ. Μετά την συνοκορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία προσπαθούμε να επηρεάσουμε την έρευνα, τις εθνικές επενδύσεις και τις αποφάσεις για την ανάπτυξη δυναμικού. Έχουμε φτιάξει αυτό τον οδικό χάρτη, μας επιτρέπει να συνεργαστούμε και μπορεί να δώσει ε, και κίνητρα για κοινά project. Από την σκοπιά της CDA, αυτός ο, αυτοί οι οδικοί χάρτες ε, έχουν και τεράστιες πληροφορίες ε, που μπορεί να ενημερώσει για, το, για τη διαδικασία ανάπτυξης δυναμικού της CDA, ε, ως συμπλήρωμα της βάσει δεδομένων συνεργατικού τύπου τη Κονταμπά, ε, που είναι και των ανοιχτών πηγών ενημέρωση. Τώρα θα ήθελα να σα ενημερώσω για την δουλειά που κάνουμε πάνω σε αυτή την ε, συνεργατική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων που λέγεται Κονταμπά ε, συγκεντρώνει πληροφορίες για πολλές χιλιάδες σχέδια, προγράμματα και ενεργοποιημένου δυναμικού ε, δυνατοτήτων στα κράτη-μέλη. Από τις ε, πληροφορίες που λάβαμε, ε, η ETA χρησιμοποίησε πάνω από 160 τέτοιες ευκαιρίες για ανάπτυξη σημαντικού αμυντικού δυναμικού και για κρατικές προμήθειες γενικής χρήσης. Αυτό ε, μας επιτρέπει να συντονιστούμε και με τους συναδέλφους του ΝΑΤΟ. Επίσης, ε, ο οργανισμός διευκολύνει την ε, αλληλεπίδραση ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προωθεί τα συμφέροντα ε, τα συμφέροντα αμυντικά σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Λόγω τη ε, εγκύτητά μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η EDA μπορεί να δώσει και σημαντικέ ευκαιρίε ε, για το ΝΑΤΟ. Παράδειγμα, το σχάρι το παράδειγμα του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, το ΣΕΖΑΡ. Θα έχει τεράστια επίπτωση στι αμυντικέ υποθέσει. Ε, θα έχει το μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη. Θα έχουμε πάνω από 2.000 μαχητικά αεροσκάφη 800 ε, μεταγωγικά αεροσκάφη και 2.600 ελικόπτερα. Με κάποιες, ε, βάσει κάποιες το κόστος του ΣΕΖΑΡ για το, στο στρατιωτικό σκέλος θα είναι μέχρι 4 δισεκατομμύρια. Και αυτό θα επηρεάσει και το ΝΑΤΟ. Κυρίω ε, την αεροπορία και τα συστήματα ελέγχου. Η EDA βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να γεφυρώσει ε, ε, τη σχέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΝΑΤΟ και θα μπορούσε επίσης και το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει το ΣΕΖΑΡ και να έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει ανησυχίε του στο EDA. Θα ήθελα τώρα να σας εξηγήσω άλλη μια φορά ότι αλλάζουν τα δεδομένα και δεν πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς. Ε, Ούτω ή άλλω και τα κράτη-μέλη μα ζητάνε όλο και περισσότερο να αντισταθμίσουμε την εδαφική άμυνα με δυναμικό διαχείριση κρίσεων και να αναπτύξουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τον υβριδικό πόλεμο. Ε, η αμυντική συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το ΝΑΤΟ. Είμαστε σε μια ε, εποχή αυξανόμενων απειλών και αύξηση του... των δαπανών για την άμυνα ή του προπολογισμού για την άμυνα. Αν δεν συνεργαστούμε τώρα, πότε θα συνεργαστούμε. Φυσικά ο δρόμο είναι μακρύ και πρέπει να μάθουμε πολλά ημένα από του ΔΕ. Αλλά κινούμαστε προ σωστή κατεύθυνση. Ακόμα μια φορά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μα δίνετε ε, να σα παρουσιάσουμε μαζί με τον ανώτατο συμμαχικό διοικητή τις συντονισμένες προσπάθειες που κάνουμε για την ανάπτυξη του στρατιωτικού δυναμικού. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας. Thank you very much. Κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στήσω τώρα από το στρατηγό Μερσιέ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. τα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Ντομέκ, κύριε και κύριοι. Είναι τιμή μου που έχω αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Με την παρουσία και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και να ζητήσω να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και συνάφεια μεταξύ του οργανισμού μας. Πριν από ένα μήνα, σε μια στρατιωτική επιτροπή όπου με κάλεσαν να μιλήσω, είπα ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι πια θέμα επιλογής, αλλά θέμα βούλησης. Πιστεύω δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά το να στηρίξουμε τις αρμοδιότητες και των δύο οργανισμών και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους περισμένους πόρους. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια παρατήρηση ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τις απαραίτητες, ε, τα ποιοτικά στοιχεία συμπληρωματικότητα για να αντιμετωπίσουν τις υψηλέ προκλήσεις του 20ου και το δυναμικό περιβάλλον του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα τώρα για τις θετικές μας ικανότητες να υπογραμμίσω το γιατί εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε περαιτέρω. Θα περιγράψω τους έξι κύριους τομείς δράσης ώστε να διαμορφώσουμε το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια. Και θα μιλήσω για τον υποστηρικτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του ACT όσον αφορά αυτό το σχέδιο ώστε να τηρηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι και του ΝΑΤΟ και της Ένωσης. Να παραθέσω καταρχάς την κυρία Μογκερίνη που είπε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ρυθμός αλλαγής θα επιταχυνθεί, θα Αντιμετωπίζουμε λοιπόν περισσότερες απειλές και προκλήσεις στο μέλλον. Όπως βλέπουμε σήμερα, στα ανατολικά και στα νότια μας υπάρχει ένας συνδυασμός όλων των απειλών που συμβάλλουν στην περαιτέρω περιπλοκότητα όσον αφορά το περιβάλλον ασφάλειας. Πράγματι νομίζω ότι εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή όπου η ρυθμίση και η επίλυση των συγκρούσεων απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ένωσης μπορέσει να βοηθήσει συμμάχους, εταίρους, χώρες να προκαταβάλουν τις κρίσεις και να αντιδρούν έγκαιρα και συνολικά, χωρίς να ξαφνιάζονται στρατηγικά. Αυτό με οδηγεί στο τρίτο μου σημείο, δηλαδή οι στρατιωτικές μας ικανότητες θα πρέπει να προσαρμόζονται αντιστοίχως για να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό αποτροπής σήμερα και στο μέλλον. Πράγματι, με την ομάδα μου έχουμε εντοπίσει έξι τομείς όπου θα μπορούσαμε να δράσουμε αντίστοιχα και να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις οποιαδήποτε στιγμή. Αυτοί οι τομείς όμως δεν είναι αποκλειστικοί του ΝΑΤΟ και μάλιστα προσφέρουν ευκαιρίες για αυξημένη συνεργασία και μπορούν να μας βοηθήσουν στο να διαμορφώσουμε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ συμμάχων χωρών και των οργανισμών μας. Καταρχάς, οι μελλοντικέ δράσεις και επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μια νέα ανθεκτικότητα και αντίστοιχες δομές και αρχιτεκτονικές ηγεσία που θα πρέπει να ευθυμεγραμμίζονται με όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και να βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διεθνών οργανισμών. Επίσης θα πρέπει να μας επιτρέπουν μια καλύτερη ανάπτυξη στρατηγικής συνειδητοποίηση ώστε να αντιμετωπίζουμε τα πρώιμα μηνύματα μιας κρίσης και να αποδίδουμε αρμοδιότητες. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν καλά αυτά τα σενάρια θέλουμε μια νέα προσέγγιση η οποία δεν θα βασίζεται σε μυστικές πληροφορίες αλλά σε ανοιχτές πηγές οι οποίες όπου χρειάζεται θα συμπληρώνονται με στοιχεία εμπιστευτικά. Και αυτό ακριβώς εδώ μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαστεί επίσης μια νέα εκπαίδευση η οποία θα προβλέπει ακριβώς αυτό το νέο περίπλοκο περιβάλλον σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ανέφερε η κυρία Μογκερίνη ώστε να αναπτυχθούν κοινέ συντονισμένες επιχειρήσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ένωση. Είχαμε αυτή την πιστοποίηση που προέρχεται από την ομάδα του Βίζεγκρατ και κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα τρίτο τομέα είναι η εταιρική σχέση. Θα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο διαδραστικότητας αν θέλουμε ακριβώς να αποφεληθούμε από την πραγματομοσύνη των περιφερειακών μας συμμάχων και να πετύχουμε σταθερότητα και να έχουμε σημαντική, σημαντικά αποτελέσματα στις επιχείρησεις μας στο ΝΑΤΟ αναπτύσσουμε ε, κάποιους οδικούς χάρτες για τους εταίρους μας που αποβλέπουν στην χάραξη στόχων διαδραστικότητας και στην απλούστευση και εξυγχρονισμό των διαφόρων πρωτοβουλειών που αναπτύσσουν οι εταίροι μας. Τα διάφορα modules με αυτούς τους οδικούς χάρτες θα μπορούσαν να προσφέρουν λοιπόν μια νέα μορφή συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την, αποφυγή επικαλύψεων. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε νέες προσεγγίσεις καινοτόμε όσον αφορά την επιμελητία και τη βιωσιμότητα. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία αρρωγή και στη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πολιτική επιμελητία και στρατιωτική επιμελητία σε ένα βιώσιμο περιβάλλον και σε τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ενδιαφέρουσε προοπτικέ. Η δυνατότητα ανταπόκριση τη στρατιωτική μα ικανότητα εξ, επίση εξαρτάται από το ανθρώπινό μα κεφάλαιο. Το ΝΑΤΟ και η Ένωση έχουν πιστοποιήσει πολλά κέντρα αριστείας και εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την απαραίτητη στάση για να αντιμετωπίσουμε τις πολλές νέες προκλήσεις. Και πάλι εδώ η στενή συνεργασία θα επιτρέψει στους οργανισμούς μας να ωφεληθούν από όλες αυτές τις γνώσεις. Και τέλος, θα πρέπει να εντοπίσουμε τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα δυνάμεων για το μέλλον, ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε όλες τις προβλέψιμες απειλές. Υπάρχει κάποια αρχική όθηση, η οποία θα πρέπει να διέπει όλους τους οργανισμούς μας σε επίπεδο ασφάλειας και αμοιβαία συνεργασία και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται αυτή τη στιγμή για ένα προπαρασκευαστικό σχέδιο έρευνας αυτό στον ε, στρατιωτικό τομέα θα μπορούσε να είναι καταλητική σημασίας και θα μπορούσε να αποδεχτεί πάρα πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα των διαδικασιών σχεδιασμού μας. Θα μπορούσαμε επίσης να διευρύνουμε το διάλογο μας με έθνη ώστε να λάβουμε γνώση των μακρόπνων σχεδίων τους και να τα ενσωματώσουμε στο δικό μας σχεδιασμό. Αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερη συνάφεια και συνέχεια των απαιτήσεων για την ικανότητα που έχουμε εμείς, ώστε να αντιμετωπίσουμε και να προσεγγίσουμε νέες διεθνείς πρωτοβουλίες, ώστε να ωφεληθούν και οι δύο οργανισμοί μας. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν στο επόμενο φόρουμ ΝΑΤΟ Βιομηχανίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Άμυνας θα διοργανώσει μια τήσια διάσκεψη στις 9 και 10 Νοέμβρη του 2016 εδώ στις Βρυξέλλες. Για τη συμβολή τώρα της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, αυτό με οδηγεί και στο τελευταίο μου σημείο. Η στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΣΥΤ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας είναι απαραίτητη και νομίζω συζητιέται σε επίπεδο αυτών των δύο οργανισμών. Ήδη πολλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω του απαραίτητου συγχρονισμού των πρωτοβουλειών μεταξύ ΝΑΤΟ και Ένωσης για τα σύνορα και τον έλεγχό τους. Το ΝΑΤΟ διερευνά αυτή τη στιγμή το πώς τα μη επανδρομένα θα μπορούσαν να ενταχθούν ακριβώς αυτή την ε, αρχιτεκτονική που προτίθεται να εφαρμόσει και ακολουθώντας τις ε, προδιαγραφές που αφορούν και τον Ευρωπαϊκό Ενίο Χώρο, τον ουρανό ώστε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα και τα στρατικά και τα πολιτικά δίκτυα. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί θα μπορούσαν συνεχώ να διευκολύνουν την ανάπτυξη μελλοντική στρατική ικανότητα, υποστηρίζοντα καινοτομία και αποφεύγοντα βεβαίω τι περιττέ επικαλύψει. Υπάρχει ανάγκη για κοινέ καινοτομίε, για, την για τον εντοπισμό των αναγκών και για την κάλυψη αυτών των κενών σε επίπεδο εθνικών ή πολυεθνικών πρωτοβουλειών. Νομίζω ότι αυτή η καινοτομία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όχι μόνο τις διαθέσιμες τεχνολογίες μέσω των διαθέσιμων εργαλείων με πλατφόρμες κλπ. Αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κατάλληλα και τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία. Και η γνώση και τα δίκτυα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα θα μπορούσαν να συμβάλλουν ακριβώ στην καλύτερη γνώση και στην καινοτομία όσον αφορά την, τον πολιτικό τομέα. Οι οργανισμοί μας λοιπόν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον συγχρονισμό των εθνικών δράσεων περιλαμβανομένων και των δράσεων των ΙΠΑ ώστε να πετύχουμε υψηλότερο επίπεδο διαδραστικότητας, διαλειτουργικότητας στο μέλλον. Τέλος, θα έλεγα ότι η δουλειά μας για την προετοιμασία του μέλλοντος ήδη έχει ξεκινήσει. Εναπόκειται σε εμά να διασφαλίσουμε το ότι οι οργανισμοί μας θα εμπλακούν. Και όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά βούλησης. Η διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ευρώπη εξαρτάται από αυτή ακριβώς την συνεργασία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι οργανισμοί μας ήδη έχουν ξεκινήσει να συνεργάζονται και προτίθενται να συμβάλλουν σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας στους ερχόμενους μήνες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Και τώρα ε, ξεκινάμε τη συζήτηση. κυρία Ίνες Αγιάλα Σάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για αυτό το πνεύμα συνεργασίας των δύο οργανώσεων που είναι σημαντικές για μας. Και είναι και σημαντική και η προσπάθεια συνεργασίας. Να ρωτήσω το εξής. Κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Πριν από λίγο καιρό ε, πήγαμε στο Γενικό Στρατηγείο, ε, ε, στην Ιταλία, Στρατηγείο για την Επιχείρηση Σοφία. Λίγο πριν ληφθεί η απόφαση να σας επιφορτήσουν, εσάς από τον, να, να επιφορτήσουν μάλλον τον ΝΑΤΟ, να ελέγχει τη Μεσόγειο στα νερά κοντά στην Τουρκία, στο Αιγαίο δηλαδή. Θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο συνεργάστηκαν οι δύο δυνάμεις στα πλαίσια της επιχείρησης Σοφία. Είχαν την εντολή να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να αποφευθούν τα ναυάγια, να σωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν θύματα των διακινητών. Και τώρα περιμένουμε το πράσινο φως για να πλησιάσουμε ε, τις ακτές της Λιβύης εν αναμονή μιας σταθερής κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αν μπορείτε να μου πείτε κάποια στοιχεία για αυτή την επιχείρηση Σοφία. Ίσως δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα αλλά αν μου δώσετε κάποια στοιχεία, ε, μπορώ να καταλάβω πιο συγκεκριμένα με ποιον τρόπο μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν οι προσπάθειες των δύο οργανώσεων. Είδαμε και στα πλαίσια της επιχείρησης επίσης Αταλάντη, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία στα ευρωπαϊκά νερά, για να το πω έτσι, ή και σε μεικτά ύδατα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λιγάκι έτσι με πιο συγκεκριμένους όρους αυτή τη συνεργασία. Thank you. Uh, ε, ευχαριστώ, ο κύριος Τζέφρι Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντοτε χαρά μας να φιλοξενούμε αξιωματούχους των, του ΝΑΤΟ και τον κύριο Ντόμεκ. Προφανώς η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πληγεί. Γιατί ορισμένες φορές είναι σαν να ε, ε, ζούμε στο δικό μας ε, κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά οι Αμερικάνοι επιμένουν στο ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στα, στο κόστος που έχει η εξασφάλιση της, ασφα, της ασφαλειάς μας. Προφανώς δεν είναι περίεργο αυτό, αλλά η απάντηση σε αυτό δεν είναι να δημιουργηθούν ξεχωριστές ευρωπαϊκές ε, αμυντικές δομές. Αντίθετα, θα έπρεπε να επικεντρώνουμε στο πώς θα μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε την συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Οι δύο οργανώσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό ακριβώς τα ίδια κράτη-μέλη. Αλλά ε, υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται εδώ στην Ευρώπη οι οποίες αποκλείουν τον, Καναδό, τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείες. 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη και του ΝΑΤΟ όλοι οι βασικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Τι, για τι πράγμα μιλάμε, κοινέ επιχειρήσεις, είμαστε σοβαροί. Αφού πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, γιατί έχουμε δύο στόλους για τις επιχειρήσεις μας στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Μα είναι δυνατόν. Είχαμε δύο στόλους στην, στην Αδριατική. όταν επιβάλαμε το εμπάργο κατά της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Υπήρχε ο στόλος του ΝΑΤΟ και μετά κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα ε, και είπε ότι όχι θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκός ο στόλος. Και έτσι είχαμε δύο στόλους. Τα ίδια πλοία από τα ίδια ναυτικά που σχημάτιζαν δύο στόλους και τελούσαν υπό διαφορετικό πολιτικό πολιτική καθοδήγηση και μέχρι και οι Γάλλοι συνήλθαν και κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ανοησίες. Γι' αυτό, όταν έχουμε αυτές τις ε, συναντήσεις, μιλάμε λίγο με αυτόν τον και καλυμμένο τρόπο και κανείς δεν λέει την αλήθεια, κανείς δεν φαίνεται να έχει το θάρρος να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Φυσικά, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας ικανότητες, το καλύτερο που θα μπορούσε να πάθει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ήταν να αυτοδιαλυθεί και να διαχυθεί στο ΝΑΤΟ. Μιλάμε για εναρμόνιση, εξυγχρονισμό, τυποποίηση. Μα το πιο σημαντικό από όλα τα πράγματα είναι οι Ευρωπαίοι, ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τον σύμμαχό μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διαλειτουργικότητα. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε διαλειτουργικοί εμείς μεταξύ μας και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν αυτή την ικανότητα. Αλλά δεν χρειάζεται να δημιουργήσει κανείς δύο ξεχωριστές οργανώσεις και μετά να δει πώς θα συνεργάζονται, αφού πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους. Μα είναι δυνατόν, γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτό. Και αν θυμηθούμε λίγο το 1998 και κατηγορώ τον ε, Βρετανό Πρωθυπουργό, ε, τον Μπλερ, τον τότε Πρωθυπουργό, που για δικούς του λόγους επέτρεψε και συμφώνησε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια δική της αμυντική ικανότητα, ξεχωριστή. Επρόκειτο για ανοησία και τρέλα. Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν συζητούνται αυτά τα θέματα εκεί, προσπαθεί πάντοτε να ε, δημιουργηθούν περισσότερες ικανότητες. Είναι ένας τρόπος για να παρακινήσουν τους, τους ε, Ευρωπαίους να κάνουν κάποιες κινήσεις. Ενώ στην, στην Ήπειρο στην ε, υπηρετική Ευρώπη, το θέμα που φαίνεται να απασχολεί τους αρμοδίους είναι πώς θα αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές αμυντικές ε, ικανότητες. Και παρά τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη Βρετανία και το γεγονός ότι σε μια εβδομάδα ο Βρετανικός λαός θα κληθεί να ε, αποφασίσει αν θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Τα δύο ζητήματα, τα κύρια ζητήματα είναι η οικονομία και η μετανάστευση. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα που υποβόσκει στη συζήτηση και είναι ο Ευρωπαϊκός στρατός. Όλοι λένε ότι κανείς δεν θέλει Ευρωπαϊκό στρατό και ο συντηρητικός ε, πρωθυπουργός της Βρετανίας σε κάθε περίπτωση ασκήσει βέτο αν έρθει τέτοια συζήτηση. Μα τίποτα άλλο δεν θα βοηθούσε και δεν θα χαροποιούσε περισσότερο τον κύριο ε, Πούτιν από αυτόν τον διαχωρισμό των δυνάμεων ε, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει επιτέλους να συνέλθουμε και να δούμε τι ακριβώς συζητείτε. Όλη αυτή η συζήτηση έχει έναν δηλητηριώδη τοξικό χαρακτήρα σε σχέση με το δημοψήφισμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η υπεράσπιση της ελευθερίας μας περνά μέσα από το ΝΑΤΟ και εκεί θα πρέπει να, κατευθύνουμε τους πόρους μας. Όλα τα άλλα είναι ανοησίες περί ολοκλήρωσης της Ευρώπης και για αυτό το πράγμα είμαι βέβαιος ότι θα το απορρίψουν οι Βρετανοί και υποψιάζομαι ότι και πολλοί άλλοι λαοί αντίστοιχη στάση θα τηρούσαν που μεταξύ αυτών βεβαίως και οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν απορρίψει κάθε συνθήκη που έχει τεθεί σε ψηφοφορία. Κανείς λοιπόν δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ας σταματήσουμε αυτές τις ανοησίες για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμενας και την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει το ένα και τις καινοτομίε και τις βιομηχανίες. Δεν χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε συλλογικά έργα άμυνας και συλλογικές επιχειρήσεις. Είχαμε πολύ επιτυχημένα τεχνολογικά προγράμματα και έργα χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Θεό λοιπόν. Ας επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι, διέρχεται πολύ επικίνδυνους καιρούς. Έχουμε μπροστά μας τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ξέρετε ότι θα μολυνθεί το κλίμα από την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σηκώσει τη δική της σημαία εκεί. Θα υπάρχουν παράγραφοι και στην τελική ανακοίνωση που θα λένε πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά είναι βλακίες. Και αυτό που εύχομαι είναι ότι όταν συνέλθει αυτή η σύνοδος, οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί θα μιλήσουν για το ΝΑΤΟ και για τίποτα άλλο. Αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμπίνε Λόζινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κάποιες πολύ γενικές σκέψεις θα σας εκφράσω εγώ. Με συγκεκριμένες προτάσεις όμως. Η πολιτική μου ομάδα πάντοτε τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια πολιτική οργάνωση αποκλειστικά μη στρατιωτική. Για κάποιον λοιπόν που δεν έχει στρατιωτική εκπαίδευση, είναι πάντοτε δύσκολο να φανταστεί κάτι τέτοιο. Ο κύριος Βαν Όρντεν ανεφέρθηκε σε αυτή την επικάλυψη ευρωπαϊκών και νατοικών στρατευμάτων Εγώ θα ήθελα να μου πείτε κάποια στοιχεία, να μου πείτε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, πώς θα μπορούσε να, τι μορφή θα μπορούσε να είχε μια ε, επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών ε, στρατευμάτων και των νατοικών. Ποια θα είναι ακριβώς η μορφή αυτής της συνεργασίας θα είναι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ή μεταξύ επιμέρους ομάδων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ ή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ποια ακριβώς θα είναι η μορφή. Επίσης, όσον αφορά τον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, ποια είναι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Task Force της με το Stratcom CIA το επιχειρησιακό κέντρο στη Ρήγα. Ευχαριστώ. Και τώρα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές μας να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους τέθηκαν και στη συνέχεια θα κάνουμε έναν δεύτερο γύρο συζήτησης. Με τη σειρά, με την ίδια σειρά Πρώτα ο κύριος Ντόμε και στη συνέχεια ο στρατηγό Μερισχέ. Ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο ερώτημα που έθεσε η κυρία Γιάλα που ε, υπερβαίνει τις δικές μου αρμοδιότητες γιατί έχει έναν επιχειρησιακό χαρακτήρα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όπως είπα και στην παρέμβασή μου ότι οι δύο επιχειρήσεις παραμένουν επί του παρόντος ξεχωριστές. Και το μόνο ε, πράγμα που παραμένει σαφές, όπως είπε και η υπατή εκπρόσωπος, είναι ότι θα ζητήσουμε υποστήριξη όσον αφορά την επιτήρηση της νέας επιχείρησης στην ε, Σόφια. Ξέρετε ότι όλα αυτά αποτελούν τμήμα μιας πολύ ευαίσθητης ισορροπίας που έχει επιτευχθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω στα άλλα δύο ερωτήματα, ιδίως εκείνα του, του κύριου Βαν Όρντεν. Γνωρίζω ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες πριν από το δημοψήφισμα και γίνονται πολλές συζητήσεις. Νομίζω ότι αυτό που δεν θα πρέπει να κάνουμε είναι να υπεραπλουστεύουμε την κατάσταση. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε, ακόμη και αν και ακόμη και όταν μιλούμε για τους ε, υπερατλαντικούς μας συμμάχους, μας έχουν πει πολλές φορές ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει με τις δικές της δυνάμεις την ασφάλειά της. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρώπη θα πρέπει να το εξασφαλίσει αυτό. Επίσης θεωρώ ότι είναι υπεραπλουστευτικό το να πει κανείς ότι χρειαζόμαστε μόνο το ΝΑΤΟ και σας διαβεβαιώ δεν πρόκειται. Το ΝΑΤΟ δεν είναι κάποιος ε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση στον ε, στο ΝΑΤΟ να καταστρέψουμε αυτό που γίνεται στο, στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Εγώ δούλεψα 10 χρόνια στο, στο ΝΑΤΟ υπό τον κύριο Σολάνα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι χωρίς μια ικανή Ευρώπη που θα μπορεί να αναλαμβάνει τις αμυντικές της ευθύνες, δεν θα υπάρχει ούτε ΝΑΤΟ. Το είδαμε και τώρα στο θέμα της μετανάστευσης. Πλέον τα ζητήματα που απασχολούν ε, τις οργανώσεις μας δεν είναι μόνο μη στρατιωτικά. Αντιθέτως, ας μην υπεροπλουστεύουμε τα πράγματα. Το ίδιο αφορά και την προστασία των ε, πολιτών μας στην ε, δική μας, στα δικά μας, στο δικό μας έδαφος με τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις, επιθέσεις που έγιναν στη Γαλλία και στο Βέλγιο, στο Βέλγιο. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να απαντηθούν, δεν θα μπορούσαν να δοθούν απάντηση σε αυτά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μόνο. Και μετά να περάσω στο θέμα του EDA που συζητείτε και έχει έναν διτό χαρακτήρα. Το πρώτο θέμα είναι να αναπτυχθούν ικανότητες των κρατών μελών ανεξαρτήτως από το πού θα χρησιμοποιηθούν. Ο ΙΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνώς. Δεν συζητούμε ποια ακριβώς θα είναι η χρήση αυτών των ικανοτήτων. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που χρειάζεται εμείς να κάνουμε είναι να προωθούμε και να ασκούμε πίεση για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, γιατί μόνο μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θα ήταν μεγάλο στρατηγικό σφάλμα να μην επιμείνουμε στην ε, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Γιατί αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες ικανότητες να ε, υλοποιούμε επιχειρήσεις που χρειάζονται, που είναι αναγκαίες για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Φυσικά. Δεν υπάρχει καν, καμία, κανένας διαχωρισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ούτε κάποια πρόθεση να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Αντιθέτως, εμείς και στους δύο οργανισμούς προσπαθούμε να υπερβούμε τους ε, περιορισμούς που υπάρχουν να αξιοποιήσουμε με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους μας και να αποφύγουμε τυχόν επικαλύψεις. Uh, να προσθέσω αυτά που είπε ο Σάφος. από δύο διαφορετικές σκοπιές να κάνω την παρέμβασή μου για τους οργανισμούς μας και τους στόχους τους. Έχουμε λοιπόν τους οργανισμούς μας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας. Αλλά στην πράξη, στην πράξη, όταν είπα προηγουμένως ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, αυτό που εννοούσα είναι ότι σήμερα έχουμε μία σχέση μεταξύ κρίσεων από ό,τι παλαιότερα. Το είδαμε αυτό στο ΝΑΤΟ, επειδή ακόμα βασίζουμε την σταδική μας δουλειά σε έννοιες του 2010, δηλαδή συλλεκτική άμυνα, συνεργατική ασφάλεια, διαχείριση κρίσεων. Αυτός ο πυρήνας αρμοδιοτήτων στο παρελθόν ήταν χωριστός. Γινόταν χωριστά όλα αυτά. Αυτό πια δεν ισχύει βέβαια. Αν λοιπόν έχουμε μια κρίση, ας πούμε, σε μια χώρα της Βαλτικής, με τη Ρωσία, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε προβλήματα στη Συρία, στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ναγκόνο Καραμπάχ. Όλες αυτές λοιπόν ε, κρίσεις αελοσχετίζονται και επειδή ισχύει αυτό, απαιτούν μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ αυτού του πυρήνα που τις ε, αντιμετωπίζει και του συντονισμού με τους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί οι κρίσεις δεν είναι μεμονωμένες πια. Αυτό λοιπόν ισχύει και κατά κάποιο τρόπο περιπλέκει τη δουλειά μας. Αλλά τουλάχιστον το καλό είναι ότι αυτό που κάναμε στο Αιγαίο και στην επιχείρηση Σόφια αποδεικνύει ότι μπορούμε να συντονίσουμε σωστά τις προσπάθειές μας και πιστεύω για το μέλλον ότι θα χρειαστεί να καθορίσουμε αρχές πάνω στις οποίες θα βασίζονται οι δικαιοδοσίε και οι αρμοδιότητες των διεθνών μας οργανισμών. Να δούμε πώς θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με την διαχείριση των επιχειρήσεών μας. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας αυτό που κάναμε το, στο παρελθόν, είχαμε διαφορετικές επιχειρήσεις, με διαφορετικό επικεφαλής ε, Ένωσης, ΝΑΤΟ, άλλο οργανισμό κτλ. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και των οργανισμών μας. Αν κοιτάξουμε τώρα τα διάφορα ευρυδικά σενάρια, ευρυδικά σενάρια που έχουμε κάποια κατόφλια για κάποιες κρίσεις, τι θα συμβεί. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε τοποθέτηση δυνάμεων υπό ηγεσία ΝΑΤΟ, κάποιες δυνάμεις υπό εθνική, εθνικές, ε, εθνική ηγεσία ή ηγεσία άλλων οργανισμών. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να τα συμπτύξουμε. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Να δούμε καταρχάς τι γίνεται με τις πληροφορίες. Δηλαδή, να υπάρχει στρατηγική γνώση η οποία δεν θα βασίζεται σε απόρριτες πληροφορίε, ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να εντοπίσουμε νωρίτερα ένα ευεργετικό σενάριο. Οι προσπάθειες μας λοιπόν θα πρέπει να συνίστανται στο να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στον τομέα της συνεργασία μεταξύ των οργανισμών μας. Και αυτό που είπα όταν κλάκεται και διαδικασία δημιουργία ικανότητας, αλλά πηγαίνει και παραπέρα αφορά το μακρόπνο σχεδιασμό. Και κάνοντας το αυτό, θα πρέπει να ενσωματώσουμε και την πτυχή της συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, που είναι πολύ σημαντικός ε, παράγοντας, και να γίνεται με την διαλειτουργικότητα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις στις επιχειρήσεις μας και θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι καλύτερες δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες οργανωτικά. Αυτό αφορά και τα πρότυπα που αναπτύσσουμε τα στρατιωτικά στο ΝΑΤΟ, αλλά και τους πολιτικούς κανονισμούς ή αυτά που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Θα πρέπει πάντως οπωσδήποτε να συνδυάζονται οι προσπαθίες μας. Και συμφωνώ και πάλι ότι η δουλειά μας είναι περίπλοκη γιατί έχουμε να κάνουμε με τόσα έθνη, 20 έθνη και διεθνείς οργανισμούς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι στο δικό μας επίπεδο ώστε να συντονιστεί καλά η δουλειά μας. Γι' αυτό ακριβώς και η κοινή δήλωση που θα γίνει στη Βαρσοβία είναι πολύ καλή, πολύ θετική. Η, η Βαρσοβία είναι η επόμενη φάση μας. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα ενισχύσει την σχέση μας και το δεσμό μας με την αντιμετώπιση, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ε, κρίσεις και τη συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών. Για την τρίτη ερώτηση που μου θέσατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθαρά πολιτικός οργανισμός, έχει και στρατηγικές αρμοδιότητες. Πώς συντονιζόμαστε λοιπόν. Καταρχάς, αυτός ο συνδεσμός μπορεί να γίνει με διάφορες επιχειρήσεις. Το ζωτικό σημείο εδώ και πάλι είναι η διαλειτουργικότητα όλων των δράσεών μας και για αυτή την διαλειτουργικότητα θα πρέπει να ακολουθήσουμε βεβαίω αυτή που ήδη ισχύει στα πρότυπα του ΝΑΤΟ αλλά και των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και χρησιμοποιείται μάλιστα και τώρα από πολλές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός ευρωατλαντικής περιοχής. Καθορίζουμε λοιπόν κάποια πρότυπα στο ΝΑΤΟ τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό ακριβώ είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα συστήματα των εθνικών στρατηγίων θα πρέπει να είναι σε επίπεδο αρχής διαλειτουργικά. Γιατί όλα τα συστήματα αναπτύσσονται ανεξάρτητα Έχουμε λοιπόν την άποψη αυτή τη στιγμή προτύπων μέσω δικτύωση. Το καλό είναι ότι οι Αμερικανοί ε, δέχτηκαν τα δικά μας τα στάντα, τα πρότυπα. το αποδέχτηκαν αυτό και αποφάσισαν να συνεργαστούν μαζί μας. Και η τελευταία χώρα που επισήμως ε, συμφώνησε να χρησιμοποιήσει αυτά τα πρότυπα είναι η Ζηλανδία. Αυτό είναι θετικό. Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αναπτυχθούμε ώστε να πετύχουμε αυτή τη διαλειτουργικότητα και να μην περιοριστούμε μόνο στον ευρωατλαντικό χώρο. Το είδαμε και στο παράδειγμα της Συρίας αυτό για το συντονισμό. Τώρα για τη στρατηγική, την επικοινωνιακή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και αυτή ακριβώς είναι η αξία του κέντρου αριστείας που αναπτύσσουμε. Το αρχηγείο μου είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση, την πιστοποίηση του ΝΑΤΟ αυτών των κέντρων αριστείας. Παρ' αυτά, αυτά τα κέντρα αριστείας αποτελούν εθνικά κέντρα. Δηλαδή, πιστοποιούνται από το ΝΑΤΟ ή άλλους οργανισμούς, αλλά είναι εθνικά κέντρα, τα οποία, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να συντονίσουν πάρα πολλά. Να είναι δηλαδή πολύ πιο ανοιχτά από ότι αν θα ήταν καθαρά τμήμα του ΝΑΤΟ, αποκλειστικά του ΝΑΤΟ. Τώρα για τη στρατηγική και τις αρμοδιότητες. Έχουμε άλλο ένα κέντρο αριστείας για θέματα κυβερνοχώρου στην Εστονία. Αυτά λοιπόν τα κέντρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους οργανισμούς μας και νομίζω αποτελούν οδηγούς που καθοδηγούν δηλαδή το συντονισμό μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στην δήλωση της Βασοβίας, της διάσκεψης κορυφής, Ένωσης ΝΑΤΟ θα αναφέρουμε το συντονισμό σε σχέση με τα ευρυντικά σενάρια. Θα αναπτύσσουμε επίσης εχειρίδια σενάριων και τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας για το πώς μπορούμε να συντονιστούμε για πρακτικά ζητήματα. Γιατί βεβαίω εντάξει, εμεί προσπαθούμε σε ρεαλιστικό καθημερινό επίπεδο να συντονιζόμαστε πάντα. Thank you, General. Uh, I kindly ask... Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Σκεφτείτε, σας παρακαλώ, οι υπόλοιποι τις επόμενες ερωτήσεις, όσο εγώ θα παρεμβαίνω. Άκουσα τον Τζέφρι Βαν και θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω μετά τα δικά του σχόλια για το γενικό θέμα της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που ασχολείται με μία πλειάδα από θέματα. Και σε όλους αυτούς τους τομείς με τους οποίους ασχολείται θέλει να πετύχει απτά αποτελέσματα. Προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στους στόχους που έχει σε διάφορους τομείς. Η ασφάλεια είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Και όταν μιλάμε για επίτευξη ισορροπίας, βλέπουμε, το βλέπουμε ξεκάθαρα ε, στην απόφαση του Jean-Claude Juncker να πάει στην Αγία Πετρούπολη. Για κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απειλή της Ρωσίας, η προσάρτηση μιας ε, εθνικά κυρίαρχης ε, χώρας, είναι άμεση φυσική απειλή. Απειλή την ύπαρξή τους. Μετά παίρνουμε διάφορες αποφάσεις λόγω οικονομικών παραμέτρων όμως. Και αγνοούμε το θέμα της ίδιας της ύπαρξης. Στη δική μου την περιοχή, εμείς προσπαθούμε να είμαστε ένα αξιόπιστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπ' την έννοια στρέφουμε τα μάτια ε, στο ΝΑΤΟ, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα εξασφαλίσει, το ΝΑΤΟ θα εξασφαλίσει την ασφάλειά μας. Όταν ήμουν εθνική βουλευτής, μας ενημέρωσαν εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ. Και πήγαινα και στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όταν ήμουν εκεί στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ παρούσα ως εθνική βουλευτή τη ε, Πολωνίας, άκουγα εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για την ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, ατζέντα για τα θέματα ασφάλειας, την προετοιμασία για τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Επομένω, μετά από όλα αυτά που σα είπα εν είδη εισαγωγής, έχω τρει ερωτήσει. Καταρχά ποια είναι η αντίληψη για τι απειλέ ε, για την ασφάλεια της Ευρώπης. Γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε την, μια κοινή αντίληψη για την ασφάλεια ή τις απειλές στην ασφάλειά μας, ούτω ώστε να αναπτύξουμε το κατάλληλο δυναμικό, τις κατάλληλες ικανότητες. Γιατί το δυναμικό αυτό ακολουθεί μετά από τον προσδιορισμό των προκλήσεων ή απειλών και σχεδιάζεται κατόπιν του προσδιορισμού αυτού. Ποια είναι η ακριβής έννοια της συμπληρωματικότητας των δύο οργανώσεων. Η ανώτατη συμμαχική διοίκηση πώς βλέπει αυτή τη συμπληρωματικότητα και πώς τη βλέπει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Είναι δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ακούσω και τους δύο κυρίους, τι άποψη έχουν. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή τους επίσης για την Τουρκία και την Ουκρανία και τη δυνατότητα συμπληρωματικής δράση απέναντι στην Τουρκία και στην Ουκρανία. κυρία Γιάλα Σέντερ. Ακόμα μια φορά θέλω να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Βανόρντεν, πρέπει να πω ότι αυτά που λέει δεν βοηθούν καθόλου την ε, δουλειά της Επιτροπής. Εγώ έκανα με κάθε έτσι ειλικρίνεια και αφέλεια, έκανα μια ερώτηση στους κυρίους. Εσείς κάνατε και μια παρέμβαση, ας πούμε ένα φιλιππικό βγάλατε. Δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνετε εδώ. Όταν εμείς οι Ισπανοί κάνουμε εκστρατεία, κάνουμε εκστρατεία. Αλλά το να ερχόσαστε εδώ πέρα και να κάνετε εκστρατεία κυριολεκτικά σε αυτή την επιτροπή ε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν νομίζω ότι είναι ο τόπο ο κατάλληλο. Κάνω την ίδια εκστρατεία τα τελευταία 17 χρόνια, λέει ο κ. Βανόρντεν. Θα σα δώσω τον λόγο αργότερα, κ. Βανόρντεν. Κυρία Γιάλα Σέντερ, σα παρακαλώ. Όχι διάλογο. Εγώ τον άκουσα με κάθε σεβασμό. Παρότι θα ήθελα και εγώ να τον διακόψω, δεν το έκανα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ, α πούμε, στη χώρα μου και μάλιστα στην πόλη μου είχαμε αμερικανικέ βάσει. Έτσι. Και μα τα λέτε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, συνεργαστήκαμε πολύ καλά ε, με τον ΝΑΤΟ. Πώς μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη είναι ε, εγωιστές, ε, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι εγωίστριες, ε, γιατί η Ευρώπη είναι εγωιστής. συνεργαστήκαμε θαυμάσια με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις, ε, ιστορικά στοιχεία, πολιτισμοί στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και τώρα αρχίζει, τώρα ακριβώς που αρχίζει, ε, μία προσπάθεια έτσι διαλόγου για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας. Δεν μπορείτε εσείς να τα βλέπετε τόσο απλουστευτικά, ότι υπάρχει μόνο μία δύναμη και τίποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Εμείς, οι ευρωπαϊκές χώρες, έπρεπε να αναπτύξουμε τη δική μας αντίληψη, τελείως διαφορετική από των Αμερικανών. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε ότι και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τις διαφορές τους. Άλλη κατάσταση στην Πολωνία, άλλη στην Ισπανία, άλλη στην Φιλανδία, άλλο στο Βέλγιο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό που κάναμε είναι ότι στην επιχείρηση Αταλάντα δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε ε, για μια καινούργια επιχείρηση με διαφορετικές εντολές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον να καταλάβουν οι πολίτες πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο οργανώσεις. Και στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο περίπλοκα πράγματα. Δεν μπορεί να έχουμε μία διοίκηση, ένα είναι ο αρχηγό, α πούμε, και όλοι οι άλλοι πακούν. όπως έγινε στη, Ρώμη, που ήρθε ένας βρετανό μάλιστα στρατιωτικό και μας εξήγησε πώς αναπτύσσεται μια πολύ ε, περίπλοκη επιχείρηση και μάλιστα μια επιχείρηση η οποία άλλαζε συν το χρόνο, άλλαζαν τα δεδομένα τη δηλαδή, ενώ είχε ξεκινήσει στην πορεία. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Η ίδια η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές χώρε, διαφορετικές αντιλήψει για το ότι είναι απειλή επίσης. Αλλά τέλος πάντων, επιτέλους, κάτι κινείται. Κάτι κινείται, ούτω ώστε και η Ευρώπη επιτέλους να λάβει τι ευθύνε τη. Νομίζω ότι πρέπει καταρχάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει μια συνένεση. Γιατί εκεί θα δημιουργούν και ευκαιρίε και για την, να τον αμυντικό κλάδο, την αμυντική βιομηχανία, τον τομέα αυτό. Και θα δημιουργηθούν ε, και θέσει απασχόληση. Ούτω ή άλλω, ε, όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνονται και στον αμυντικό τομέα στην Ευρώπη, τις βλέπουμε πολύ θετικό μάτι και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία. Πρέπει να συνεργαστούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να κάποια στιγμή αναλάβουμε και εμεί τι ιστορικέ μα ευθύνε. Είναι περίπλοκη αυτή η πορεία, όπω είναι περίπλοκη και η πραγματικότητα. Είναι τελείως δια... Έχουμε δύο διαφορετικέ αντιλήψει για την άμυνα εδώ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έχουμε από τη μία τις ευρωπαϊκές απειλέ και από την άλλη τι παγκόσμιε απειλέ. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε μία συνολική θεώρηση. Αυτά. Mm-hmm. Uh, Κύριε Βαν Όρντεν, θέλετε το λόγο. Κύριε Στετίνα. τα τότε... Είμαι ευρωβουλευτής εδώ και δύο χρόνια και φαίνεται, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ευρωβουλευτών. Η μία ομάδα που προέρχεται από, την, από τις παλαιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός και αφετέρου η ομάδα των Ευρωβουλευτών που ε, προέρχεται από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Και η δεύτερη αυτή ομάδα έχει μια εντελώς διαφορετική ιστορική εμπειρία από την πρώτη ομάδα. Η πρόεδρος αναφέρθηκε ότι η ρωσική απειλή έπειτα από τις επιθέσεις στην Κρυμαία και στο Ντομπάς είναι εξαιρετικά υψηλή και όσοι προερχόμαστε από πρώην σοσιαλιστικές χώρες βλέπουμε πραγματικά αυτόν τον κίνδυνο και σας καλούμε παρακαλώ ακούστε μας στρατηγέ εγώ πρόσφατα βρέθηκα στο Ντομπάς και μίλησα και με αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων της ε, Ουκρανίας και μίλησα και με τάγματα εθελοντών. που συμμετείχαν σε διενέξεις, σε συγκρούσεις στον Ντονμπάς και στο Λουγκάνσκ και μας είπαν ότι δεν έχουν πυρομαχικά, δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν όπλα και χρειάζονται την υποστήριξή μας. Ο, ο πόλεμος είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Έχουν πεθάνει 10.000 άνθρωποι Και εγώ αναρωτιέμαι, είμαστε διατεθειμένοι ως μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούμε σε αυτές τις εκκλήσεις για βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να, κλείσουμε τα σύνορα, να κλείσουν τα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οι στρατιώτες που βρίσκονται εκεί πολεμούν εδώ και δύο χρόνια και Λένε όλοι ότι αν κλείσουν τα σύνορα, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μέσα σε ένα μήνα. Οπότε το ερώτημά μου είναι, τι μπορεί να γίνει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάριο Κιούρεκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Βλέποντας αυτήν την ε, πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη του ΝΑΤΟ. Καμία από αυτές τις χώρες δεν έγινε πρώτα ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια του ΝΑΤΟ. Μπορεί να έγινε σε διαφορετική χρονική στιγμή, αλλά για όλες τις χώρες μας πρώτα ναι, ενταχθήκαμε στο ΝΑΤΟ και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όσον αφορά την ασφάλεια σε χώρες όπως η Πολωνία, οι Βαλτικέ χώρες, η Τσεχία ή ακόμη και η Βρετανία, εμείς όταν, αντιλαμβανόμαστε την, όταν σκεφτόμαστε την ε, ασφάλεια, εννοούμε τη συνεργασία μέσω του ΝΑΤΟ και η συμπληρωματικότητα για εμάς πρέπει να λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτή τη διάσταση. Και ένα δεύτερο θεμελιώδες για μένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένωση κρατών ή είναι κάτι διαφορετικό. Αν είμαστε ένωση κυρίαρχων κρατών, τότε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και πράγματα τα οποία γίνονται μόνο σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω τα κράτη-μέλη της Ένωσης να ε, συνεργάζονται σε θέματα ασφάλειας με συμπληρωματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Αλλά στο ΝΑΤΟ είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί είναι εκείνοι που επομίζονται το μεγαλύτερο τίμημα αυτού του νέου ψυχρού πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη παρά το γεγονός ότι οι συγκρούσεις δεν γίνονται στην ε, Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να γίνουμε πιο ενεργοί και όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και όσον αφορά την καταπολέμηση ε, της προπαγάνδας της Ρωσίας, η οποία κατευθύνεται ενάντια στην Ευρώπη και όχι ενάντια στη ΣΥΠΑ. Και κάτι τελευταίο. Το ΝΑΤΟ βεβαίως έχει ως βασικό του στόχο την ε, άμυνα, τη στρατιωτική άμυνα. Οποιαδήποτε άλλη δράση του μπορεί να είναι μόνο συμπληρωματική. Πρόληψη, για παράδειγμα. Η πρόληψη μπορεί βεβαίως να ενισχυθεί και να γίνεται κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωενωσιακό επίπεδο. Θυμόμαστε όλη την έκκληση του Προέδρου Ποροσέγκο, την οποία δεν ε, έκανε μόνο προς τη δική μας Επιτροπή, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αποσταλεί μια ειδική αποστολή στην, ε, στην Ουκρανία, μια εκτελεστική αποστολή η οποία θα έχει ως καθήκον την ε, επιτήρηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας του Μίνσκ. Δυστυχώς τίποτα δεν συνέβη. Δεν μιλώ για αστυνομική αποστολή, αλλά μια αποστολή η οποία θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Όταν μιλούμε για συμπληρωματικότητα, θα πρέπει επίσης να εξετάζουμε και συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά πολιτικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, Στην ε, δική μου χώρα, πολλοί βουλευτές αλλά και ευρωβουλευτές επικρίνουν την επιχείρηση Ανακόντα. Ενώ στην πραγματικότητα, στόχος αυτής της επιχείρησης ήταν να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι ακούστηκαν τέτοιες φωνές. Και αν κοιτάξει κανείς πραγματικές λύσεις που μπορούν να δοθούν που θα ενισχύσουν και την ε, δέσμευσή μας στην ασφάλεια και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η βασική μας συμβολή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των στρατευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί διαφορετικά τελικά θα καταλήξουμε κάθε κράτος μέλος να χαράσει μια δική του πολιτική. Γιατί ακριβώς τα, κράτη, τα περισσότερα κράτη αντιλαμβάνονται την άμυνα ως έναν κύριο τομέα του ΝΑΤΟ. Πρόεδρος, όσον αφορά την Ουκρανία και τις αποστολές που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο έδαφος αυτής της χώρας, αυτά τα θέματα λοιπόν έχουν συζητηθεί πολλάκις στην Επιτροπή μας. Και όποτε συζητούμε το θέμα της Ουκρανίας, πάντοτε κάνουμε σχετικές εκκλήσεις και πάντοτε έχουμε και προσκεκλημένους από την Ουκρανία. Είμαστε λοιπόν μία από εκείνες τις επιτροπές που πραγματικά ε, συμμετέχουν δραστήρια και ενεργά στην προώθηση τέτοιου είδους εκκλήσεων. Λοιπόν, πρωτού δώσω το λόγο και πάλι στους ομιλητές, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Μούρεκ που σχετίζεται με την ε, ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει το ΝΑΤΟ σε αυτόν τον τομέα είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θέλουμε δηλαδή να διατηρήσουμε ένα προφίλ ότι οι οργανώσεις μας θέλουν να προωθήσουν την τεχνολογική καινοτομία. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ποια είναι λοιπόν η κατεύθυνση στο συγκεκριμένο θέμα που έχει χαραχθεί. Πρώτα θα δώσω το λόγο, τον, ε, το λόγο στον κύριο Ντόμε και στη συνέχεια στον κύριο Μερσιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανερχόμαστε στο θέμα της αντίληψης της απειλής. Στην θεώρηση για την απειλή, η ανάλυση των κινδύνων των απειλών, ουσιαστικά είναι κάτι το κοινό και στις δύο οργανώσεις. Ή την ανάλυση της μίας οργάνωσης την παίρνει η άλλη. Δεν είναι αυτή ανάλυση, αυτή καθεαυτή που μετράει για να λάβεις ε, δράση. Το θέμα είναι η αντίληψη που έχει κανείς για αυτή την απειλή. Και μην ξεχνάμε επίσης ε, και το θέμα των γειτόνων μας. Το είδαμε στην επιχείρηση για τη Λιβύη. Είχαμε διαφορετικές ευαισθησίες, κατα... καταφέραμε όμως να τις αντιμετωπίσουμε γιατί υπήρχε συμπληρωματικότητα στη δράση. Ε, φυσικά, αν θέλαμε να δεν θα πρέπει να είμαστε και απλουστευτικοί υπερβολικά. Πρέπει να σας πω, για, για τη συλλογική άμυνα, το ΝΑΤΟ είναι η πρώτη επιλογή, αλλά δεν είναι η μόνη λύση που πρέπει να σκεφτόμαστε σήμερα πια. Και τώρα πάμε στο τι σημαίνει αυτή η συμπληρωματικότητα στην πράξη. Το σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε μόνο τα αμυντικά θέματα σήμερα. Πρέπει να σκεφτούμε την ασφάλεια και την άμυνα συνολικά των πολιτών σήμερα. Αν δείτε ότι γίνεται, γίνεται τι γίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω της μετανάστευση. Και το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία εντολή σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Αλλά έχει κάποιο δυναμικό, κάποιες ικανότητες που μπορούν να βοηθήσουν δυναμικό για τη Frontex και εκεί η Frontex μπορεί να διαθέσει ό,τι πληροφορίες έχει. Η επιχείρηση στο Αιγαίο θα μπορούσε να έχει δώσει περισσότερους καρπούς αν ήμασταν σε διαφορετικό πλαίσιο. Αλλά υπάρχει μια συνεισφορά εκεί και του ΝΑΤΟ ε, και, της, και της άλλης οργάνωσης, δηλαδή υπάρχουν καρποί από τη συνεργασία. Τώρα, οι συνολικές απειλές για την Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό απορρέουν από την κατάσταση στη Συρία. Ε, εκεί δεν χρησιμοποιήθηκε το ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα ποιο είναι οι τρομοκρατικές απειλές ε, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό. Ίσως και εδώ θα πρέπει να δούμε τη συμπληρωματικότητα των μέσων. Δηλαδή τι μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θα ήταν ανόητο να μην χρησιμοποιήσουμε την πιο σφαιρική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριλαμβάνει και την ασφάλεια και την άμυνα, αλλά και όλο το δυναμικό του ΝΑΤΟ. Στην EDA, στη δική μου, στο δικό μου οργανισμό, αμυντικό οργανισμό, να σας δώσω δύο-τρία παραδείγματα ε, πάνω σε αυτά που κάνουμε. Που τα κάνουμε εμεί, αλλά το ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται να τα κάνει ή δεν μπορεί να τα κάνει, αλλά πρέπει να τα κάνει η Ευρώπη. Μιλήσαμε και στο παρελθόν για έλλειψη ε, ανεφοδιασμού σε καύσιμα αέρος-αέρος στην, Εμεί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Και το αντιμετωπίσαμε σε επιχειρήσει που δεν ήταν υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και χρειάστηκε να ζητήσουμε από του Αμερικανού να μα εξασφαλίσουν αυτό το δυναμικό. Όταν λοιπόν ε, μιλάμε για αμυντικέ επενδύσει, θα πρέπει να δούμε και πού, θα επενδύσουμε, σε τι είδου ε, δυναμικό ε, και δυνατότητε πρέπει να επενδύσουμε όπου δεν τι έχουμε ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι επίση να αυξήσουμε μόνο τον προπολογισμό, να τον αυξήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε καλά. Καταρχά είναι οι τεχνολογίε ε, ανάπτυξη και δεύτερον ε, ε, επενδύσει σε προμήθειε. Όχι μόνο σε προσωπικό, σε προμήθειε, σε αγορέ. Δεν έχει νόημα να αυξάνουμε το προσωπικό, να προσλαμβάνουμε κόσμο αν δεν υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό, αν δεν έχουμε τι κατάλληλε προμήθειε. Ε, έχουμε τώρα για τον, τον ανεφοδιασμό αέρος-αέρος έχουμε τα τάγκερ των Αμερικανών και εξασφαλίζουμε άδειε ε, για να ε, ανεφοδιάζουμε τα μαχητικά μας αεροσκάφη ε, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση. Γιατί άμα προσπαθήσουμε να ανεφοδιάσουμε τα αεροσκάφη αυτά αφού ξεκινήσει η επιχείρηση, χάλασε η ιστορία, χάλασε η επιχείρηση. Ε, επίσης, υπάρχει νομοθεσία και κανονισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, στο επίπεδο του REACH, που ρυθμίζει τις χημικές ε, ουσίες του εξοπλισμού. Αυτό έχει τεράστια επίπτωση σε όλη την αμυντική βιομηχανία ε, και στην αμερικανική βιομηχανία επίσης και για τον εξοπλισμό που οι Αμερικανοί σύμμαχοι βάζουν και βγάζουν από την, στην Ευρώπη. σε περίπτωση που υπάρξει ή τον εξοπλισμό που θα βάλουμε ας πούμε, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκό α, έδαφος. Πώς εξασφαλίζουμε την αρμόνιση. Την... Εμείς, το ΝΑΤΟ δεν το κάνει αυτό, έτσι. Εμεί λαμβάνουμε υπόψη τι, έχει το ΝΑΤΟ, τι μα διαθέτει το ΝΑΤΟ κτλ. Και εμεί εξασφαλίζουμε την εναρμόνιση. Τώρα, για την προπασκευαστική δράση ε, που θα ενταχθεί στον προπολογισμό, ε, ή μάλλον που θα καταβληθεί υπομορφή πρόταση τη Κομισιόν, θα υποβληθεί στην υπομορφή πρόταση τη Κομισιόν και θα έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου προ εξέταση. Το βασικό είναι να είμαστε αλληλολειτουργικοί κτλ. Δεν μπορούμε εμεί να χαλαρώσουμε, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία ε, και να περιμένουμε του Αμερικανού. Ε, Εάν δεν ανασκουμποθούμε τώρα, θα χάσουμε το τρένο και δεν θα μπορούμε στρατηγικά και επιχειρησιακά να παίξουμε κάποιο ρόλο και να σταθούμε στο πλευρό των Αμερικανών. Και να έρθω σε ένα τελευταίο παράδειγμα. Μιλούσατε για τις ε, χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. που βρισκόταν πίσω από το σιδηρό παραπέτα, το σιδηρό παραπέτασμα. Εμείς στον οργανισμό μου κάναμε μια προσπάθεια καλύτερης ένταξης ε, του κλάδου, του αμυντικού κλάδου αυτών των χωρών στην ε, αλυσίδα ανεφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας της ε, Ευρώπη. Οι Αμερικανοί δεν είναι κάτι που θα το, θα το κάνουν αυτό. Δεν είναι στην εντολή του ΝΑΤΟ, δεν είναι προς το συμφέρον του. Ε, προ συμφέρον του, αλλά εμεί το κάνουμε στο δικό μου οργανισμό, στην EDA, στον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Ε, Επίση, αναφερθήκατε στην Τουρκία και στην Ουκρανία. Για την Τουρκία. Υπάρχει μια διοικητική ε, διευθέτηση με την EDA που έχει μπλοκαριστεί από το 2006 για την Τουρκία. Εάν προχωρήσουν διαπραγματεύσεις ε, φέτος για το θέμα της Κύπρου, ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την συμφωνία για την ε, Τουρκία. Και με την Ουκρανία έχουμε υπογράψει το Δεκέμβριο μία διοικητική ε, συμφωνία που θα μας επιτρέψει να ασχολήσουμε, για, να δουλέψουμε για τον, σε επιχειρήσεις υποστήριξης για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, και θα υποφεληθούμε ημένα από τους δε, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι δηλαδή. Στρατηγέ. Ευχαριστώ ένα συμπληρωματικό σχόλιο. Για τις απειλές. Και πώς το αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ. Εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις απειλές που προέρχονται από όλε τι πλευρές της ευρωατλαντική περιοχής. Όπως είπα προηγουμένως, συνδέονται μεταξύ τους. Το είδαμε αυτό στη Συρία και αλλού. Δεν γίνεται λοιπόν να διαχωρίζουμε τις απειλές ας πούμε, από την Ανατολή σε σχέση με απειλές από άλλα μέρη. Για την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Υπάρχει μια διαφορά στην προσέγγιση μεταξύ δύο οργανισμών μας που πρέπει να κατανοήσουμε. Στην Ένωση υπάρχει ένας κατάλογος ικανοτήτων. Στο ΝΑΤΟ δεν ακολουθούμε το ίδιο δρόμο κοιτάμε τι στόχους έχουμε, οι οποίοι χαράσσονται στις στρατηγικές στρατηγικούς οριζόντες, που ακολουθούν την πολιτική χάραξη των στόχων, η οποία μας καθοδηγεί. Είναι λοιπόν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Τώρα βρισκόμαστε στα μέσα μιας τετραετούς διαδικασίας στο ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη ικανοτήτων και σε μια φάση σχεδιασμού. Τώρα στέλνουμε στις χώρες μέλη στόχους, όχι μόνο για την ικανότητα, αλλά με συγκεκριμένους αριθμούς. Θα πρέπει μετά από κάποιο καιρό να δούμε ακριβώς κατά πόσο στα Υπουργεία Άμυνας έχουν επιτευθεί αυτοί οι στόχοι για τον αέριο ανεφοδιασμό. Το ίδιο ισχύει. Όταν εμείς λοιπόν εντοπίζουμε κενά, πάμε και κάνουμε έρευνες σε όλες τις χώρες και όταν έχουμε κάποια αποτελέσματα τα στέλνουμε σε όλους. Έχουμε ομάδες που συμμετέχουν μέλη και από τους δύο οργανισμούς μας. Το κάνουμε εν μέρη χωριστά, αλλά όχι ακριβώς, και ο ενάριος αρεφοδιασμός είδαμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας θα ήταν ο καλύτερος οργανισμός για να το προωθήσει. Είπαμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε ικανότητα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Αυτό νομίζω το καλύτερο δείγμα συνεργασίας μπορούμε να έχουμε. Τώρα, να σας πω πάλι ότι έχουμε κάποιες κοινέ δομές αλλά το κυριότερο είναι να ενθαρρύνουμε τις χώρες να αποκτήσουν υποδομές και ικανότητα ανάλογα με τους στόχους τους. Και αν αποδειχτεί καλύτερο, μπορούμε να τα κάνουμε και αλλιώς. Μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε κοινέ πρωτοβουλίε. Για την Ουκρανία έχουμε μια σοβαρή εταιρική σχέση με την Ουκρανία μέσω προγραμμάτων εταιρική σχέσης του ΝΑΤΟ. Κάνουμε πολλά με την Ουκρανία. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους. Και στο Norfolk, στο στρατηγείο μου, δεν έχουμε μόνο χώρες ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε και αξιωματικούς από την Ουκρανία που δουλεύουν. Έχουμε και πολλές πρωτοβουλίες εταιρικής σχέσης με την Ουκρανία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική γενικότερα η εταιρική μας σχέση με την Ουκρανία. για την πρόληψη. Ναι, για τη συλλογική άμυνα είναι ο καταλληλότερο οργανισμό του ΝΑΤΟ. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όμω, όμω, το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ δεν περιορίζεται στη συλλογική άμυνα μόνο. Στη Βαρσοβία αντιμετωπίζουμε δύο κυρία θέματα για τη διάσκεψη ένα πώς θα ενισχύσουμε αποτροπή και άμυνα σε σχέση με κρατικές απειλές αλλά και μη κρατικές απειλές και δεύτερον ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ να αφορά την προβολή της σταθερότητας το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολλές εταιρικές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες όπου και οι εταίροι μας θα συμμετέχουν στις δράσεις πρόληψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε όλες τις χώρες εταίρους να είναι ανθεκτικές και να αντιμετωπίσουν ε, απειλές τρομοκρατικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσης. Έχουμε από τη Μεσόγειο μέσω διαλόγου καλύτερη σχέση με αρκετέ χώρες και εκεί ακριβώς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις στις υπόλοιπε δραστηριότητε και δράσει που έχουμε με τα άλλα κράτη-μέλη. Έχει όμω το ΝΑΤΟ τεράστια ευθύνη και σε αυτόν τον τομέα επίση. Το θέμα τώρα της συμπληρωματικότητας των δύο οργανισμών μας. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση της Λιβύης θα είναι σταθερή και αν θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια επιχείρηση στην Λιβύη. Εδώ όμως έχουμε δύο διαφορετικά προβλήματα. Έχουμε καταρχάς την ανάπτυξη του ISIS, πρόβλημα τρομοκρατίας, πρόβλημα με τους πρόσφυγες, με τα σύνορα, με την οικοδόμηση της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν συνεργασία μεταξύ των οργανισμών μας. Το ΝΑΤΟ είναι ο κατάλληλο οργανισμό αν χρειαστεί να καταπολεμήσουμε, α πούμε, τους τρομοκρατικές οργανώσει, το ISIL κτλ. Υπάρχουν οι κατάλληλε διαδικασίε για την λήψη πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω είναι καταλληλότερη για κάποιε άλλε δραστηριότητε, ενδεχομένω και ο ΙΕ και κάποιες άλλες χώρες. Αυτό εννοούσα έλεγα, που έλεγα προηγουμένως ότι δεν είναι ασπρομαύρο ένωση να το αποκλειστικά δηλαδή. Αντιπαραθετικά. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αν αυτό το είχαμε κάνει και στη Λιβύη κιόλα, μετά τον πόλεμο, μετά τις μάχες εκεί, αν είχαμε λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση, δεν θα αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό νομίζω είναι και το σημείο κλειδί για το μέλλον. Και τέλος, για την τοποθέτηση δυνάμεων σε θέσεις μάχης. Βρισκόμαστε σε φάση σχεδιασμού, όπως σας έλεγα, για την ανάπτυξη δυνάμεων και την επίτευξη των στόχων μας. Θεωρώ ότι όλες οι δυνάμεις και οι ευρωπαϊκές στρατικές δυνάμεις, οι ευρωπαϊκές μονάδες θεωρούμε ότι μπορούν και αυτές να χρησιμοποιηθούν και να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ικανότητα του ΝΑΤΟ. Και αυτό ακριβώ συνδέουμε την πιστοποίηση που σας έλεγα προηγουμένως με τις μεγάλες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, όπως κάναμε το 2015. Διαφορετικά, στο εσωτερικό μιας χώρας θα υπάρχει ένας διχασμός μεταξύ δυνάμεων ΝΑΤΟ, δυνάμεων Ένωσης. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, γιατί μιλάμε πάντοτε για τις ίδιες στρατηγικές δυνάμεις. Οπότε διαφωνώ κάπως με αυτά που είπε προηγουμένως ένας ομιλητής. Για το ΕΣΥΤΗ e προσπαθούμε για το μέλλον να προκαθορίσουμε τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις και απαιτήσει για την ασφάλεια και την όσον αφορά τις μηχανίες αλλά πρέπει η βιομηχανία και το δύο πλευρών του Αταντικού να εμπλακεί. Όπως βεβαίως και η Ευρωπαϊκή σε αυτή την τόσο σημαντική δραστηριότητα, ώστε να υπάρχει η σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο μας. Και ήμουν σίγουρη από την αρχή ότι η συζήτηση θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως και αποδείχθη ότι ήταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, για τις παρεμβάσεις σας, τις πολύτιμες παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής για αυτήν την έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση που έθιξε όλα τα σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστούμε και για τις ε, πολύ ολοκληρωμένες και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σας. Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ. May I ask you to be seated? Sorry. May I ask your attention? Thank you. Next. Actual. Λοιπόν, επόμενο και τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξής μας είναι ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. μεγάλη μου χαρά υποδέχομαι και καλωσορίζω στην Επιτροπή μας ένα, μια διασημότητα της πολιτικής. Αλήθεια είναι, δεν υπερβάλλω. Υπουργό της Ισπανίας, ε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ε, είπα το εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και πρόεδρο του ευρύτερα γνωστού κέντρου ΕΣΑΝΤΕ της Μαδρίτης, κέντρου παγκόσμιας οικονομίας και γεωπολιτικής. Και το θέμα που θα συζητήσουμε είναι πώς θα τεθεί σε εφαρμογή η παγκόσμια στρατηγική προοπτικές για μια λευκή βίβλο για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις και να δώσω τον λόγο στον κύριο Χαβιέ Σολάνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που επανέρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, το οποίο επισκεπτόμουν επί δεκαετία πολύ συχνά. Τελευταία φορά που ήρθα ήταν πριν από, 20, ε, πριν από 6 χρόνια νομίζω. Έχει περάσει λοιπόν πολύ καιρό. Τα συναισθήματά μου λοιπόν είναι πολύ έντονα, είμαι συγκινημένος και χαίρομαι πολύ που μου ζητήθηκε η συνεργασία μου για να εξετάσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν τομέα που πιστεύω ότι για όλους μας είναι πολύ σημαντικό. Άμυνα και ασφάλεια σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε μια συνεχή, συνεχή μεταβολή και εξέλιξη και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομική κρίση για παράδειγμα, θα πρέπει να μην ξεχνάμε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι η ασφάλεια και η ε, άμυνα. Θέματα δηλαδή τα οποία θα πρέπει να επανέλθουν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα εδώ είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει ε, έπειτα από δύο εξελίξεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, η συνθήκη της Λισαβόνας που ανοίγει δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα και δεύτερον, η νέα στρατηγική ε, για την ασφάλεια που θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες η είπατε εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε οι σχετικές εργασίες επί μου το 2003 όταν και συνειδητοποιήσαμε ότι το τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο ε, μεταβαλόταν και έκτοτε πράγματι ε, το τοπίο έχει αλλάξει τόσο πολύ που χρειάζεται μια νέα ματιά. Άρα έχουμε αφενός τη συνθήκη της, Λισαμο... Λισαβόνας και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει και το περιεχόμενο της νέας στρατηγικής, στρατηγικής που θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω αλλά αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι το εξή. Η ιδέα είναι γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη ολοκλήρωση όσον αφορά την πολιτική άμυνα και ασφάλεια στην Ευρώπη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για ένα απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής μας. Ακριβώς διότι αυτά τα δύο στοιχεία ε, που ανέφερα, η συνθήκη της Λισαβόνας και η νέα στρατηγική για την ασφάλεια, δεν έχουν αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Και ο κόσμος περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες στον διεθνή, στην διεθνή σκακέρα και γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη μας, στην ε, γειτονιά μας, εκτός της γειτονιάς μας και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δούμε πόσο μπορούμε να αναπτύξουμε αυτά που έχουν ήδη εγκριθεί αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει λοιπόν από την ψήφιση της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ανεπαρκείς κατά τη γνώμη μου. Και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εξετάσει αυτά τα θέματα και το ενδεχόμενο σύνταξης μιας λευκής βίβλου πρέπει να εξατιστούν ε, όλα αυτά τα θέματα. Πρώτον, οι δαπάνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αυτές που είχαν ε, εξαγγελθεί και χωρίς αύξηση των δαπανών δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Υπάρχουν από το 2008 πάρα πολλές ε, προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Πάρα πολλές χρόνος και πάρα πολλές προσπάθειες κατευθύνθηκαν ε, στο πώς θα ενισχυθούν και θα αυξηθούν τα χρήματα για την οικονομία. Και έτσι ξεχάστηκαν κατά κάποιο τρόπο τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας. Και βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε χάσει κάποιες δυνατότητες και κάποιες ικανότητες που έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί στο σωστό χρόνο, το 2010, το 2011 κτλ. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, τα ξέρετε όλα αυτά, αλλά είναι εμφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την ικανότητά της να διατηρεί την παρουσία της σε μια σειρά ε, μέτωπα. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος του 2%. Πολύ λίγες χώρες, ακόμη και στους προϋπολογισμούς του 2016, κινούνται προς μια τέτοια κατεύθυνση του 2%. Οι προϋπολογισμοί μας είναι πολύ περιορισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με το επίπεδο των δαπανών που θα υπάρχει, που δεν νομίζω να είναι 2%, αλλά θα πρέπει εμείς να κοιτάξουμε πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι δεν σημειώνουμε πρόοδο στο ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η αναγκαία και η εφικτή, η επιθυμητή ε, διαλειτουργικότητα. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης, όχι θέμα χρημάτων. Πόσο θέλουμε να καταστήσουμε διαλειτουργικά τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι δεν έχουμε καταβάλει επαρκείς προσπάθειες όσον αφορά την άρση των επικαλύψεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι αποτελεσματική η χρήση των ε, πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Πολλά πρέπει να γίνουν. Και φυσικά, επειδή δεν είναι εύκολο να εξεύρει κανείς οικονομικούς πόρους, θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε και τις διαδικασίες εξοικονόμησης πόρων και χρημάτων. Νομίζω ότι οι στρατιωτικές δομές επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί στον στον μέγιστο βαθμό. Πολλά μπορούν να γίνουν εκεί και πολλά μπορούν να γίνουν και στον τομέα της συνεργασίας. Το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που θα θέλαμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και εγώ θυμάμαι ότι όταν το 2004 δημιουργήσαμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, είχαμε θέσει κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί. Η απόφαση λοιπόν, οι αποφάσεις που έλαβε ο οργανισμός αυτός το 2004 δεν έχουν τύχει της απαραίτητης υποστήριξης από τα κράτη-μέλη. Όπως βλέπετε λοιπόν, εγώ θα επικεντρωθώ ε, κυρίως σε πράγματα που έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά που δεν έχουν γίνει. Κάποια από αυτά τα θέματα σχετίζονται με χρήματα και κονδύλια, αλλά όμως ε, σχετίζονται με την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τα οικονομικά θέματα, και τα χρηματοδοτικά, αλλά νομίζω ότι το κύριο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η αποτελεσματικότερη ε, εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν την συνθήκη της Λισαβόνας. Η οποία μας δίνει μια πλειάδα από θέματα. Ε, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, προς το παρόν έχουμε αποφασίσει διάφορα να μην τα κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει, ενισχυμένη συνεργασία που είναι κλασική για όλους τους τομείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα. Και για να υπάρξει κάτι τέτοιο, χρειάζεται μια πλειοψηφία. Προς το παρόν, αυτή η πλειοψηφία δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ε, τίποτα για την ισχυμένη συνεργασία, όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά για την άμυνα και για διάφορα άλλα θέματα. Υπάρχουν για, υπάρχουν για θέματα ε, ασφάλειας και άμυνας η διαρθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ. Αυτό τι σημαίνει, ότι ένας μικρός αριθμός χωρών μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν αυτή την προκεχωρημένη συνεργασία, την ενισχυμένη συνεργασία, όπως τη λέμε, συνθήκη της Λισαβόνας. Τίποτα δεν έχει γίνει και εδώ. Έχουμε δύο δυνατότητες για να κάνουμε κάτι παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Επίσης, στον τομέα τη χρηματοδότηση, υπάρχουν πολλά, πολλά κενά, πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει. Υπάρχει ένα μηχανισμός ενισχύ, αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει Γιατί ο τρόπος που επιμεριζόμαστε τα βάρη είναι ένας τρόπος που δεν κινητοποιεί τις χώρες για να κάνουν κάτι. Αντίθετα. Γιατί όποια χώρα κινητοποιείται, ας πούμε, πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Και οι υπόλοιπε χώρε που ακολουθούν επωφελούνται χωρί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. δεν είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να δρούμε, αν θέλουμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα, έτσι. Το θέμα είναι πώς θα μοιραστεί το βάρος. Στην πραγματικότητα, λέει, θέλουμε να αποποιηθούμε το βάρος. Και όταν αποποιούμε αυτό το βάρος, τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι γίνεται τελικά. Κάτι πρέπει να γίνει προς αυτή, ε, προς αυτή την κατεύθυνση επίσης. Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες συνεργασίας για τα αμυντικά θέματα. Έχουμε τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας. Την έχει επικαλεστεί η Γαλλία. Δηλαδή, η... σε αυτή την περίπτωση, μία χώρα ε, ζητάει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν. Ε, Επίση, υπάρχει και ρήτρα αλληλεγγύη για να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μέσω τη συνθήκε και λόγω του πώ είναι διαμορφωμένο το τοπίο στα θέματα ασφάλεια και άμυνα, απαιτείται μια πολύ μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν δεν γίνει καμία αλλαγή στους κανονισμούς που έχουμε, στη συνθήκη ας πούμε. Έχουμε τη συνθήκη, έχει εγκριθεί. Θα έχουμε σύντομα μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο Έχουμε τεράστιο περιθώριο να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά που κάνουμε σήμερα, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα σε ρυθμιστικό, κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο. Δεν έχω διαβάσει 100% την παγκόσμια στρατηγική και επομένως, ε, είναι δύσκολο να τη σχολιάσω σήμερα και να πω πώς μπορούμε να τη συμπληρώσουμε. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν πράγματα τα οποία μπαίνουν στη στρατηγική και τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα τα καταστήσουμε λειτουργικά, ε, κάποια πράγματα δηλαδή επίσης που λείπουν από την παγκόσμια στρατηγική θα πρέπει να τα εντοπίσουμε και να τα εντάξουμε. Λοιπόν, εν συνεχεία πρέπει να δούμε, αφού εντοπίσουμε τα capabilities, ε, το δυναμικό δηλαδή, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Όταν δείτε τις, την κατάσταση της χώρας μας, τη χώρα μου κτλ, το θέμα της ασφάλειας είναι βασικό μέλημα. Θέλω να ε, σκεφτείτε την ασφάλεια και την άμυνα ως ένα σύνολο. Επίσης, οι επιλογές, μας που, κάνουν, οι επιλογές που κάνουμε ε, έχουν επιπτώσει σε τρίτες χώρες και αντίστροφα. Το να μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα, είτε για εντός είτε για εκτός, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω είναι η λάθος προσέγγιση. Ε, είναι ένα σύνολο το τι συμβαίνει εντός και εκτός και ξέρετε ότι όταν έχουμε προβλήματα ε, στην εσωτερική ασφάλεια, αυτά τα προβλήματα ουσιαστικά τα εισάγουμε, προέρχονται από προβλήματα στο εξωτερικό και αντίστροφα. Επομένως, θα πρέπει να βλέπουμε τα θέματα ασφάλειας και άμυνας ε, ως ένα σύνολο. Εσωτερική και εξωτερική άμυνα και ασφάλεια. Είναι ένα όλον. Αυτό είναι εκ των νόνου κάνευ. Είναι μια νέα προσέγγιση, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι που έχει συζητηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, από όλε τι χώρε έχει συζητηθεί, έχουμε κάποιες ευθύνε ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη και όταν διαβάζετε τα έγγραφα τα οποία σας παρουσίασα σήμερα. Ε, Στην συνεχεία θα πρέπει να γίνουμε πιο επιχειρησιακοί. θα πρέπει τα προγράμματα και τα μέτρα α, να τα κάνουμε, ε, να τα προωθούμε σε άλλο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή τα προωθούμε ε, με έναν όχι απλώς αργό ρυθμό, με το ρυθμό του μείον άπειρο ας πούμε, της χελώνας. Ε, φυσικά ο ρυθμός μας δεν είναι η ταχύτητα του φωτός, αλλά δεν χρειάζεται να κινούμαστε και με το ρυθμό της χελώνας ας πούμε. Ε, θα πρέπει να βρούμε το δικό μας ρυθμό, καλύτερο ρυθμό και να μην χάνουμε ούτε λεπτό, γιατί δεν μας περιμένει κανένας. Είμαστε τμήμα αυτού του πλανήτη και είμαστε μεταξύ των ηγετών αυτού του πλανήτη. Έπειτα, για την έρευνα και τεχνολογία. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ειδικά στο, στις διπλές χρήσεις. Δηλαδή κάνουμε κάτι σε ένα τομέα και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο τομέα και μπορεί να έχει επιπτώσει σε άλλο τομέα. Ή παραδείγματο χάρη στην. Κάνουμε κάτι σε βιομηχανικό τομέα, μπορεί να έχει ε, επιπτώσεις και στην ασφάλεια. Ε, επίσης, χρηματοδοτικά κίνητρα μπορεί να επηρεάσουν εταιρείε. Ε, εταιρείε οι οποίες κάνουν τεχνολογικές ε, καινοτομίες ε, και που μπορεί να επηρεάσουν το πεδίο, το, τοπίο της ασφάλειας. Αυτά που κάνουν οι εταιρείε με τη σειρά τους. Επίσης, κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου. Η ασφάλεια... Ας, ας αποκτήσουμε για την ασφάλεια και την άμυνα κάτι αντίστοιχο με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δηλαδή, οι χώρες σε αυτό το τομέα, όταν δεν σέβονται τις δεσμεύσεις τους, θα πρέπει να προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία ε, μέσω ε, μιας βαθμολόγησης που θα κάνουμε στην, στις επιδόσεις των χωρών αυτών. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε στο ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για να δούμε τι έκανε μια χώρα σε σχέση με αυτό που δεσμεύτηκε να κάνει. Και να γίνονται, να δίδονται κίνητρα μέσω εξέταση από αμοτήμου, ούτω ώστε να κινητοποιούμε τι χώρε να κάνουν περισσότερα από αυτά που κάνουν σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπει και αυτό στο εγγύ μέλλον. Ε, το, μέχρι το 2020 μέχρι το 2025 θα δούμε τι ορίζοντα θα έχει. Αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια, αυτό σας λέω, ότι πρέπει να έχουμε κάποια αναφορά, δηλαδή κάποιο σημείο αναφοράς με το οποίο θα μετράμε τις επιδόσεις, ας πούμε, με βάση το οποίο θα μετράμε το τι πετύχαμε. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συμπληρώσει τη στρατηγική της σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, θα πρέπει να έχει έναν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα καταρχάς, έξι μήνες, ας πούμε ένα χρόνο, για να βλέπει τι δεν έχει κάνει και να το συμπληρώνει. Και συνεχεία να προχωράμε από εκεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την ύπατη εκπρόσωπο να αναπτύξει μία λευκή βίβλο για την ε, εφαρμογή των στοιχείων του εγγράφου που σας παρουσίασα εγώ, υπό μορφή σχεδίου. Και να δούμε τι αντιστοιχεία υπάρχει με τα αποτέλεσματα της παγκόσμιας στρατηγικής, του Global Strategy. Η ύπατη εκπρόσωπος, νομίζω, θα πρέπει να ηγηθεί μία ομάδα ανθρώπων όπου θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Στατιωτική Επιτροπή και αφού δημιουργηθεί μία ομάδα υψηλού επίπεδου με τους υφυπουργούς άμυνας ή κάποιους ομοτήμους τους, εν σε υψηλό επίπεδο δηλαδή, και όπου τα ευρωπαϊκά κράτη και, και τα Υπουργεία Άμυνας μπορούν να εμπλέκονται για να βλέπουν τι, τι παίζεται. Επίσης, ο, γενικός ο βοηθός γενικός γραμματέας της ΚΕΠΑ θα μπορούν να εμπλέκονται. Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία, ή μάλλον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Και επίσης και το στρατιωτικό προσωπικό, οι στρατιωτικοί θα πρέπει να συνεισφέρουν για να καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα capabilities. Η ύπατη εκπρόσωπος θα συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Και κάθε στιγμή μπορούν, μπορεί κάποιος να εξετάζει τους κανόνες. Όλα αυτά σε διαβούλευση με εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον ΝΑΤΟ. Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται σε συνεργασία, σε συντονισμό ή με ενημέρωση του ΝΑΤΟ. Θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι εξάντλησα το χρόνο μου. Προσπάθησα να κάνω αυτό που μου ζητήσατε όταν με καλέσατε. Να παρουσιάσω κάποιες ιδέες με οργανωμένο τρόπο. Να εξετάσουμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας. Υπό την αιγίδα της, είπα, της εκπροσώπου. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Έχει αλλάξει το τοπίο της ασφάλειας τόσο πολύ που θα ήταν βλακώδες να μην το κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να το κάνουμε με ενεργητικότητα, με αποφασιστικότητα και ζήλο. Όλα αυτά που σας λέω είναι συμβατά με τους κανονισμούς που έχουμε σήμερα και με τη συνθήκη της Λισαβόνας, που είναι το βασικό δίκαιο με βάση το οποίο δουλεύουμε μέχρι να αλλάξει βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω το έγγραφο αυτό να σας βοήθησε και να σας βοηθήσει στην ε, δουλειά που σας περιμένει και στη δουλειά που περιμένει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Το γράφουν οι, οι εφημερίδες κάθε μέρα στα πρωτοσέλιδα και εμείς το αντιμετωπίσουμε σαν στα ψηλά γράμματα. And, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει Πρόεδρος. να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Αν έχετε παρατηρήσεις, πείτε μου. Να πω και εγώ ότι το προηγούμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή μας ήταν συζήτηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ ΝΑΤΟ ΕΕ. είχαμε τον επικεφαλής της του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του ACT από το ΝΑΤΟ. Και ένα από τα σημεία που συζητήσαμε αφορούσε την συμπληρωματικότητα όσον αφορά τις δράσεις των δύο οργάνων. Μας είπε ο διοικητής του ACT ότι το ΝΑΤΟ σχεδιάζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και θέτοντας απαιτήσει ή προποθέσει για τα μέλη του ΝΑΤΟ, λαμβάνοντα υπόψη βέβαια μια περιφερειακή ισορροπία, χωρίς βεβαίως να εξαιρεθεί η Ευρώπη από εκεί. Μα έλεγε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος συμμαχός μας, η ΕΠΑ, επιθυμούν να αυξηθεί ο ρόλος και η συμβολή μας στην κοινή άμυνα. Μας είπαν ότι καταρχάς θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερο οικονομικό βάρος με την αποτελεσματική και ευφυή χρήση των πόρων, των οικονομικών. και να αυξήσουν ταυτόχρονα τους στόχους αυτούς εσείς τι θεωρείτε όσον αφορά την ουσιαστική αποτελεσματικότητα της Ευρώπης και επίσης όταν μιλάμε για ανάληψη ευθυνών συχνά αυτό συνδέεται από την ανάγκη αυτονομίας. Οπότε εδώ πώς τα συνδυάζουμε τα δύο, πώς τα συμβιβάζουμε. Αυτή δηλαδή την περιφερειακή ισορροπία του ΝΑΤΟ και την αυτονομία εντός Ένωσης όσον αφορά την οικοδόμηση ικανότητας. Αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση. Και πείτε μου αν κάποιος άλλος έχει το λόγο. Θα προσπάσω να απαντήσω λέγοντας το εξής. ήμουνα γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σε δραματικές στιγμές, σε εποχές διεύρυνσης και του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και ήμουν επικεφαλής και είπα τους εκπρόσωπος για θέματα ασφάλειας. Από την προσωπική μου εμπειρία να σας πω το εξής. πρέπει να υπάρχουν πιο ολοκληρωμένες ικανότητες στην Ένωση. Αυτό είναι καλό για την Ένωση και καλό για το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα μέγιστα αν δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε αυτό το τομέα που όπως έλεγα αφορά εσωτερική εξωτερική ασφάλεια σε αμοιβαία διάδραση. Αφού γίνει λοιπόν σε επίπεδο ένωσης, μπορεί μετά να επεκταθεί στο ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι και η δέσμευση που έχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν δράσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, του διευρυμένου ΝΑΤΟ και των επιχειρήσεων της Ένωσης που ήδη έχουμε κάνει Κατά τη θητεία μου είχαμε πάνω από 30 επιχειρήσει εκτό Ένωση. Νομίζω αρκετά επιτυχή. Σταματήσαμε βέβαια να το κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι στο ΝΑΤΟ τώρα έχουμε κάποιο θέμα με την Τουρκία, αλλά και πάλι το είχαμε ρυθμίσει τότε κατά τη θητεία μου. Τέλος πάντων, αυτό που είπατε, η λέξη αυτονομία, όταν γίνεται μια αποστολή αυτόνομα από την Ένωση, λαμβάνεται η απόφαση σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Γεωγραφικά, μια περιοχή μπορεί να μην είναι η κατάλληλη για δράση από το ΝΑΤΟ. Οπότε θεωρούμε πρέπει να δούμε τις περιπτώσεις όπου το ΝΑΤΟ τέλο πάντων θέλει να δράσει αυτόνομα, οπότε η Ένωση εδώ επισέρχεται. Μπορεί να υπάρξουν λοιπόν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να δράσει όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και σημερινά παραδείγματα ή του πρόσφατου παρελθόντος ή του άμεσου μέλλοντος που μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο όπου το ΝΑΤΟ ή η δεν θέλουν να παρανεύουν. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αυτό είναι αμφίβολο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απεμπλεκόμαστε από το ΝΑΤΟ τη που η το των χωρών μελών είναι και του ΝΑΤΟ. Ω ΝΑΤΟ όμω μπορεί να μην θέλουν να δράσουν ή να παρανεύουν. Δεν λέω τίποτα μυστικό, αλλά φαντάστε ότι αυτό συζητιέται με τη ΣΥΠΑ. Σε συζητήσει, σε φόρουμ στη ΣΥΠΑ που είπα τα ίδια πράγματα που λέω και εδώ. Πριν 10 χρόνια θα είχα διαφορετική ανταπόκριση από την ανταπόκριση που έχω σήμερα. Η ΕΠΑ λοιπόν, ο πιο σημαντικός παράγοντας του ΝΑΤΟ, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν θέλει να δράσει, δεν θέλει να παρενέβει για συγκεκριμένου λόγου, οπότε πρέπει να το κάνουμε εμεί. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είμαστε σε αντίφαση, ότι αντιφάσκουμε. Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο και δεν κάνουμε τίποτα το οποίο αντιφάσκει με τον ΝΑΤΟ ή τη ΣΥΠΑ. Αυτό δεν θα ήθελα τώρα να το δραματοποιήσουμε. Και πρέπει να δούμε, να το δούμε σε σχέση με τους παγκόσμιους μας στόχους. Να μην το δραματοποιήσουμε λοιπόν, αλλά βέβαια θα υπάρξουν στιγμές όπου θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε μόνοι μας. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και πρέπει να μας είναι ένα δίδαγμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε τώρα τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Θετίνα πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σολάνα, Είπατε ότι ήσασταν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πράγματι, ήταν δύσκολη εκείνη η περίοδος. Να σας υπενθυμίσω τι είχε πει τότε ο πρόεδρος Βάσλαβ Χάβελ για την ε, επέμβαση στο Κόσοβο. Είχε πει ότι πιστεύω ότι η επιχείρηση στο Κόσοβο. δεν είχαν ως κίνητρο την αποκόμιση κάποιου ωφέλους, κάποιου κέρδους. Ήταν ανθρωπιστική και μόνο οι λόγοι. Θα ήθελα λοιπόν μιας και μιλούμε σήμερα για το ΝΑΤΟ και το μέλλον του. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και να αναλύουμε το παρελθόν ε, του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορέσουμε να χαράξουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο το μέλλον του οργανισμού. Ο κύριος Τζέφρι Βαν Όρντεν. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Σολάνα. Είπατε για το Πέσκο. Ποιος θα αναλάβει τα ενία σε αυτή τη διαδικασία. Και πείτε μας λίγο ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα του να ακολουθήσουμε ε, το Πέσκο. Η κυρία Λόζιν. Ευχαριστώ. Κύριε Σολάνα, εδώ, εδώ είμαι, εδώ, στα αριστερά σας. Είπατε ότι δεν έχετε διαβάσει ακόμα τη στρατηγική για την ασφάλεια. Κανείς μας δεν την έχει διαβάσει γιατί δεν υπάρχει ακόμη. Δεν έχει δημοσιευθεί. Παρ' όλα αυτά, η ύπατη εκπρόσωπος έχει εκφράσει ορισμένες στρατηγικού χαρακτήρα σκέψεις της. Εγώ έχω διαβάσει ό,τι έχει δημοσιευτεί στην, στην, ιστοσελίδα. Αν λοιπόν τώρα συζητήσουμε την εκπόνηση κάποιας λευκής βίβλου, τότε αυτές τις πολύ γενικές σκέψεις που μέχρι στιγμής έχουν εκφραστεί, το ζητούμενο θα είναι να τις μετουσιώσουμε σε συγκεκριμένες πράξεις. Και θα ήθελα να μάθω από εσάς πώς πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πράξεις και μέτρα αυτές οι γενικές σκέψεις που έχουν εκφραστεί. Προφανώς ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον είναι η συμπληρωματικότητα, δηλαδή που μπορούν να δράσουν από κοινού και συμπληρωματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και αυτό που με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο είναι πώς θα ε, μπορέσουμε τις διάφορες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Βανόρντεν. Δεν μιλούμε μόνο για στρατιωτική ικανότητα. Αυτό που διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ΝΟΑΤΟ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτική συμμαχία, αλλά διαθέτει και αρμοδιότητες σε τομεί μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Και σε αυτό, σε αυτό το θέμα νομίζω ότι αυτή η συμπληρωματικότητα ε, είναι πολύ σημαντική προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις, ε, ε, αρμοδιότητες και τις δυνατότητες των δύο οργανισμών. Επίσης, υπάρχουν διάφορα εργαλεία για την ανάπτυξη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει στα, στα χέρια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα πρέπει αυτά τα εργαλεία να ενταχθούν και να συμπεριληφθούν και στη στρατηγική για την ασφάλεια, αλλά και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και τέλος, μιλούμε πάντοτε για τη χρηματοδότηση. Και υπάρχει βεβαίως και αυτό το αίτημα από πλευράς ΝΑΤΟ για 2% αμυντικές δαπάνες στους προπολογισμούς. Δεν είναι και νέο αυτό. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε ε, αν χρειάζεται να επαναληφθεί αυτό το αίτημα. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια άμεσα για, την, ε, για τις ε, αμυντικές δαπάνες. Με βάση τη συνθήκη κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, αλλά υπάρχουν διάφορες ερμηνείες που έχουν ακουστεί. Αναφερθήκατε και στην έρευνα. Και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να ενισχυθεί και να προωθηθεί η έρευνα με ευρωπαϊκά χρήματα. Ποια είναι η γνώμη σας. Είπατε επίσης, αναφερθήκατε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, που είναι και αυτό ένα πολύ επίμαχο θέμα και στον τομέα της οικονομίας και σε ποιον βαθμό περιορίζονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, ιδίως αν επεκταθεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό εξάμεινο και στον στρατιωτικό τομέα. Φαντάζομαι ότι θα, αν κατατεθεί τέτοια πρόταση θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούν να συμβάλλουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί στους στόχους που έχουν τεθεί ώστε να ενισχυθούν τα κονδύλια και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τελικό ερώτημα. Αυτή την προοπτική μιας λευκής βίβλου ε, την έχουμε ε, μπροστά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όμως πιστεύετε εσείς ότι δεν εκπονήθηκε ποτέ αυτή η λευκή βίβλος. Σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία και ποιες δυνάμεις φρενάρουν τη σύνταξη μιας τέτοιας λευκής βίβλου. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που άλλαξα τη σειρά με την οποία παίρνουν το λόγο ε, οι πολιτικές ομάδες. Δεν ήξερα ε, ότι οι σοσιαλιστές είχαν ζητήσει το λόγο. Με συγχωρείτε. Κύριε Άννα Γκόμες, έχετε εσείς το λόγο. Ευτυχώς που ήρθε ξανά ο κύριος Σολάνα. Και ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα έγκαιρα να τον ακούσω, αλλά υπόσχομαι ότι θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον την μελέτη που μας παρουσίασε. Δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να, όχι απλά να σας καλωσορίζω, να σας θέσω και κάποια ερωτήματα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε ε, στο τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει και να δράσει ακόμα και μόνη. Και αυτό σημαίνει προετοιμασία, σημαίνει το να έχει το απαραίτητο δυναμικό, τις απαραίτητες ικανότητες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια κατάσταση στο Ιράκ, Φερρυπίν, που την, την είδα, ε, που είναι το Ιράκ μία από τις χώρες ε, τους προμαχώνες καταπολέμησης του ISIS. Κάποια κράτη-μέλη δίνουν όπλα ε, γι' αυτό, αλλά χωρίς κανένα συντονισμό. Και δεν ρωτήσαμε ποτέ, ρωτήσατε εσείς ποτέ την ε, κυρία Μογκερίνη, μάλλον ψέματα, εγώ την ρώτησα την κυρία Μογκερίνη, να, ρωτήσει, να μου πει γιατί δεν συντονίζει τα κράτη-μέλη. Και είπε ότι δεν είναι δουλειά της ε, δικής τη υπηρεσίας ε, που ασχολείται με την εξωτερική πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Επίσης, στη Λιβύη, διάφορα κράτη-μέλη εμπλέκονται, δεν το παραδέχονται, αλλά μονομερώς έχουν, αναλαμβάνουν δράσεις. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια αποστολή ΚΠΑ ακόμα και για να βοηθήσουν οι χώρες αυτές, οι ευρωπαϊκές χώρες, να οικοδομηθεί ένας στρατός εκεί, κάτι που δεν είχε ποτέ πραγματικά η χώρα αυτή, ένας ενιαίος στρατός. Θα ήταν πολύ σημαντικό για να ξεπεραστούν και τα προβλήματα που σχολείς ότι υπάρχουν η κυρία Μογκερίνη για το θέμα της ετοιμότητας. Επενδύσεις και στην έρευνα και τεχνολογία, κατάρτιση κτλ, ασφάλεια. Έχουμε ακούσει ε, κάποιες εκθέσεις ότι οι Ρώσοι έχουν τους φακέλους με μέλη του δημοκρατικού, των δημοκρατικών κομμάτων. Ε, αν μπορούν να το κάνουν σε τρίτες χώρες, μπορούν να το κάνουν παντού και στην Ευρώπη. Επίσης, πώληση όπλων από τις ε, επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, γιατί ε, μπορεί να πουλάνε και κρίσιμες υποδομές. Ε, μην ξεχνάμε επίσης ε, και συμβόλαια ε, σε επιχειρήσεις και κινέζικες κτλ. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Αρχίζουμε τουλάχιστον να συνειδητοποιούμε ότι υπολοιπόμεθα σε σχέση με το που βρισκόμαστε 10 χρόνια πριν. Και τέλο, εάν φύγει η Βρετανία, αν αυτό αποφασιστεί το δημοψήφισμα και ελπίζω όχι, αυτό σίγουρα θα είναι αρνητικό, γιατί δεν θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό εταίρος ό,τι αφορά την οικοδόμηση δυναμικού στον τομέα της ασφάλειας. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτό το κόμμα που κάνει αυτό το δημοψήφισμα είναι και το κόμμα που βάζει συνήθως τις τροχοπέδες στο τι μπορούμε να κάνουμε στη συνεργασία μας. Μιλάμε στην, για τη Βρετανία. Thank you and last in the... Τελευταία παρέμβαση σε αυτό το γύρο ερωτήσεων. Η κυρία Ινές Αγιάλα Σέντ. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ και καλωσορίζω τον κύριο Σολάνα στην Επιτροπή μας. να αναφερθώ σε δύο πολύ σημαντικά που είπε. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε, παρόπου είναι δύσκολο και δυσκολότερο στο Κοινοβούλιο και έχει καταθέσει και μία τροπολογία εγώ, για τη συγκρούση μιας υποεπιτροπής, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε όλα τα θέματα ασφάλειας εντός και εκτός. Γιατί τώρα Έχουμε νομικές βάσεις τελείως διαφορετικές, διαφορετικές προσεγγίσεις. Είμαστε υπό την αιγίδα των εξωτερικών, με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, επιφέρει επιπλοκές και κάποιες φορές τα πολύ σημαντικά δεν μπορούμε καν να τα συζητήσουμε γιατί πάνε κατευθείαν και ψηφίζονται στην εξωτερικών υποθέσεων. Μειονέκτημα αυτό. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν εσωτερικά κάποιες ανάγκες και κάποιες ικανότητες που πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό ήθελα λοιπόν εγώ να σχολιάσω. Πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να συμβάσουμε αυτά τα δύο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δώσουμε ένα κίνητρο στις χώρες μέλη Μετά το δεύτερο, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα ως κίνητρο για τη δημιουργία μιας δυναμικής ώστε να προχωρήσουν όλες οι χώρες μέλη και να μπουν σε επίπεδο κινητοποίησης. Γιατί αυτοί που κινητοποιούνται περισσότερο το κάνουν μέσω μιας εντάξει θεμητής μηχανικής πολιτικής όμως που δεν περιέχει το άλλο κομμάτι, το πολιτικό, και πρόοδου. Ενώ το πολιτικό καμιά φορά παραβλέπει είτε το στρατηγικό που έχουμε συζητήσει επαναλημμένως εδώ ή την απουσία του μηχανικού κομματιού που έχει και αυτό να κάνει με τα κίνητρα και την ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αυτό το εξάμεινο πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να προσπαθήσω να τις απαντήσω. Αλλά να πω πρώτα ότι είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω ένα πιθανό, μάλλον μια ενδεχόμενη διαδικασία για μια λευκή βίβλο. Δεν μπορώ να σας δώσω απόψεις προσωπικές για θέματα τα οποία δεν σχετίζονται με την παρουσία μου εδώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ βέβαια, αφού φαίνεται ότι σας ενδιαφέρουν και βαραίνουν οι δικές μου απόψεις αλλά το Κοινοβούλιο με κάλεσε να προσθέσει το έγγραφο, το οποίο εντάξει δεν είναι λευκή βίβλος, αλλά μια διαδικασία προς μια λευκή βίβλο. Αυτό είναι κάτι που παλιότερα ούτε καν διαδικασία δεν ήταν. Τώρα όμως υπάρχει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την Ένωση. Επιτρέψτε μου όμως να είμαι πολύ προσεκτικός για αυτά που θα πω. Έχω προσωπικέ απόψει, οι οποίε όμω δεν αφορούν το λόγο τη παρουσία εδώ σήμερα. Είναι αλήθεια ότι το παρελθόν είναι τμήμα του μέλλοντος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και να γίνει στο παρελθόν, εντάξει, να το πάρουμε υπόψη μας, αλλά το δίδαγμα, το δίδαγμα του παρελθόντος είναι το να δούμε το μέλλον και να μην συνεχίσουμε να κοιτάμε το παρελθόν. Νομίζω ότι οι δράσεις μας στο παρελθόν ήταν σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένη περιοχή της γειτονιάς μας και ήταν η πρώτη φορά που επικράτεια της Ένωσης περιλάμβανε ένα πόλεμο, τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι η απάντηση που χρειαζόταν δόθηκε. Δόθηκε σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους, με τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς, τον ΟΗΕ. Θυμάμαι το τον κύριο Κόφη Ανάν που είχε αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες και συνεργάστηκε στενά μαζί μας. Είχαμε λοιπόν μια πολύ καλή, πολύ ευφυή συνεργασία. Και όταν έγινε γενικός γραμματέας, ήρθε στην Ευρώπη, έκανε κάποιες συνδεύξεις τύπου, οπότε με συνεργασία λοιπόν του ΟΗΕ αντιμετωπίσαμε την κατάσταση στα Βαλκάνια. αυτό το δίδαγμα. Η προεκβολή όμως των δαγμάτων πρέπει να γίνει ευθυώς, γιατί η κατάσταση σήμερα δεν είναι ίδια με αυτή πριν κάποιο καιρό στη γειτονιά μας. Πέρασε πολλή χρόνος. Έχουν συμβεί διάφορα. Και να μην κάνουμε προεκβολές γραμμικές. Το συμβάντο δηλαδή τη δεκαετία του 90 στον 21ο αιώνα. Εντάξει, λίγα χρόνια έχουν περάσει τώρα ε, από τότε που μπήκε ο 21ος, αλλά τόσο ο 21 ο αλλα τελο παντων βρισκομαστε στον 21ο, τι να κάνουμε. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τη συνεργασία. Αυτό δεν είπατε. Η ΠΕΣΚΟ. Η μη ΔΣ Η μόνιμη δομένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ. Όχι, έχει λάθος έκανα. Για την Πέσκο μιλάγατε, για τη Μούδου Σου. Νομίζω ότι η ενισχυμένη συνεργασία και η δομημένη συνεργασία είναι κάτι το οποίο κατά δική μου την άποψη είναι σημαντικό και θα ήταν έξυπνο, ευφυές, πιστεύω, να περιληφθεί στη διάσκεψη γιατί νομίζω προέρχεται από την στρατηγική της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω για κάποια θέματα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει σε κάποιες χώρες να προχωρήσουν πέραν αυτών που είναι υποχρεωτικά και αν θέλουν να το κάνουν. Και βέβαια να είναι ανοιχτή η δυνατότητα συμμετοχή και των υπολείπων. Η ενισχυμένη συνεργασία δεν είναι κάτι το κλειστό, είναι κάτι το ανοιχτό. Και οι χώρες που συμμετέχουν θα πρέπει βέβαια να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι δεν ισχύουν για όλους. Η δομημένη και η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να αφορά αυτούς που το επιθυμούν. Όσοι λοιπόν μπορούν και θέλουν, να το κάνουν. Αλλά όπως και η Ευρωζώνη δεν περιλαμβάνει, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους όσους αυτούς θέλουν δεν θα ήταν κακό να δούμε αυτές τις δύο κλασικές περιπτώσεις που συνδέονται ακριβώς με την ουσία των κρατών εθνών και την δυνατότητα συνεργασία τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι η ιδέα που είχαμε κατά νου όταν ξεκίνησε το Σύνταγμα. Και τελικά συμφωνήθηκε η περίληψη, η παραμονή αυτή τη ιδέα στην συνθήκη τη Λισαβόνα. Νομίζω είναι κάτι το θετικό όμω, το οποίο μπορεί να έχει καταληκτικέ επιπτώσει. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να γίνει, να γίνει. Η κατάλυση με και επιστήμονα είναι κάτι που μου αρέσει. Γιατί χωρί την κατάλυση πολλά πράγματα θα γινόταν. Ε? Αυτή λοιπόν η καταληκτική επίδραση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό λοιπόν το είδο ε, καταλυτικής επίπτωσης είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας επιτρέψει να ωφεληθούμε όσοι δηλαδή θέλουν να μπορούν να το κάνουν έστω και με ετεροχρονισμό. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Δεν κομίζω γλάφκας, αλλά είναι δική μου άποψη και τέλο πάντων βασίζεται και σε αυτά που έγιναν στα πλαίσια της συνθήκης κλπ. Δεν μπορώ να πω λοιπόν τίποτα άλλο. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό στην δομημένη συνεργασία. Ιδιαίτερα τώρα που μπορούμε να κάνουμε την παραβολή με την Νομισματική Ένωση, που είναι άλλη μια μορφή δομημένη συνεργασίας. Πάντως, Πρόεδρε, για την ε, ικανότητα είναι σημαντικό αυτό που είπατε και νομίζω αφορά και αυτό που είπα. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ μέσα-έξω, εσωτερικού-εξωτερικού. Νομίζω τον κόσμο σήμερα θα πρέπει να τον δούμε με μια διαφορετική προοπτική. Αν κοιτάξουμε τις χώρες έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά αν σκεφτούμε τις χώρες έθνη, τότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ένωση. Κατά πάσα πιθανότητα το κράτος έθνος περιλαμβάνει βεβαίως τη διοίκηση στην εσωτερική. Ε, η αστυνομία, ο νόμος, η δικαιοσύνη κτλ. κτλ. Αυτό χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των πολιτών και για τη χρήση των στρατιωτών εκτό συνόρων. Έτσι. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να, το, είναι να το αντιστρέψουμε αυτό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εκτό όχι μόνο του στρα, στρατιωτικού, αλλά και στοιχεία που χρησιμοποιούμε για την ασφάλεια των πολιτών μα. Π.χ. σε επιχειρήσει χρησιμοποιήσαμε, α πούμε, στοιχεία τη αστυνομία, τη δικαιοσύνη, των πραγμάτων που δεν σχετίζονται ιστορικά με την εξωτερική μας δράση και αφορούν τη διακυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό νομίζω λοιπόν είναι πολύ σημαντική διάκριση τη σήμερα ημέρα. Στο τέλος του 20ου και αρχές του 21ου αυτά που κάναμε δεν ήταν μόνο στρατιωτικά, ήταν στρατιωτικά συν, πλάς, λέει ο Πρόεδρος. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι στρατιωτικά μείον, δηλαδή ενισχυμένη αστυνομική και ελαφρύ light στρατιωτική. Κοσφοπέδιο και σε άλλα μέρη τέλος πάντων. Αυτό που κάναμε ας πούμε στο Κοσφοπέδιο ήταν μια αστυνομική αποστολή. Δεν ήταν στρατιωτική, βοηθούσε την ασφάλεια στη χώρα. Αυτά είναι λοιπόν πράγματα που τέλος πάντων θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Όταν εγώ μιλάω για μια συνέχεια, για μια συνεκτικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία καλούμε ασφάλεια με την ευρεία έννοια, όχι μόνο με την παραδοσιακή στρατιωτική έννοια. Τώρα, στους δρόμους του Παρισιού, των Βρυξελών, θα βρείτε τέλο πάντων στρατιωτικούς οι οποίοι ασχολούνται με τη εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Αυτό δεν το βλέπαμε παλιά στις δημοκρατικές χώρες. Τώρα χρειάστηκε να το κάνουμε επειδή είχαμε μια απειλή τέτοιας φύσης. Έχουμε λοιπόν πράγματα τα οποία είναι καινούργια, που δεν είχαμε φανταστεί παλαιότερα. Και αντίστροφα, πρέπει να προβλέψουμε πράγματα για εξωτερικές δράσεις που δεν είχαμε προβλέψει στο παρελθόν. Αυτή είναι η νέα κατάσταση. Και μεγάλες χώρες ακόμα, η εκεί να προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Και η Ευρωπαϊκή λοιπόν θα πρέπει και αυτή να το κάνει και για περισσότερους λόγους, γιατί έχουμε μια διάσταση πιο περίπλοκη. Πρέπει να το κάνουμε λοιπόν εμείς. Αυτό κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, να το συζητήσουμε, επειδή αποτελεί την ουσία των βασικών αργών που βιώνουμε. Οι διανέξεις τι αφορούν. Τα εδάφη, τις χώρες, τον κυβερνοχώρο. Δεν θα μπορείτε να στείλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στρατιώτες στο ίντερνετ, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Πρέπει ούτως ή άλλως να προστατεύσετε τη χώρα σας, ας πούμε, από κυβερνοεπιθέσεις. Οπότε όταν αντιμετωπίζεται α πούμε μια επίθεση στα πνευματικά δικαιώματα. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείτε τα ίδια εργαλεία, τις ίδιες λύσεις. σε κάποιε περιπτώσει πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ίδια εργαλεία όπω η προστασία μια σημαντική επιχείρηση από επιβουλέ. Αυτή λοιπόν είναι η κυρία συζήτηση που πρέπει να γίνει μεταξύ μα και νομίζω ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ που θα χρειαστεί πολύ καιρός ώστε να συντονιστούμε στις δράσεις μας ώστε αυτές να είναι επίκαιρε με τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, αν είχαμε χρόνο θα το είχαμε κάνει. Πάντως, για να απαντήσω στην ερώτηση σας, ναι, προβλέπω την ύπαρξη δράσεων οι οποίες προϋποθέτουν, όπως είπα, τη συμμετοχή στοιχείων όπως αστυνομία, δικαιοσύνη κτλ. και που εκπροσωπούν τη δικιά μας υπόσταση τελικά των Ευρωπαίων. Εκπροσωπεύουν τις δικές μας ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες δεν είναι μόνο θεωρητικές αλλά και εφαρμόσιμες. Αυτό είναι και το οποίο μας διακρίνει. Και είμαι περήφανος που ανήκω σε ένα οργανισμό που έχει θέσει αυτούς ως στόχους όχι μόνο για μας, αλλά παγκοσμίως. Τώρα, για τη χρηματοδότηση. Όπως είπα, στην αρχή είναι περίπλοκο αυτό. Και καμιά φορά οδηγεί στην ε, αποθάρρυνση των χωρών για δράση. Γιατί αυτός που δρά πληρώνει. Και είναι λοιπόν μια αποτροπή για δράση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μηχανισμούς οι οποίοι θα είναι πιο ισορροπημένοι. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα γίνει αυτό συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τρόπους. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας ταχύς οικονομικός μηχανισμός και δίκαιος να υπογραμμίσω και τη λέξη ταχύς. Όταν μιλάμε για θέματα ασφαλείας, ο χρόνος είναι κάτι το ζωτικό. Αν λοιπόν δεν είστε έτοιμοι να δράσετε ταχαίως, τότε καλύτερα να μην δράσετε καθόλου. Γιατί θα γίνει ζημιά. Οπότε για τον μηχανισμό, γιατί κάποιος ρώτησε για τον μηχανισμό, είναι αλήθεια ότι οι μηχανισμοί είναι δυσκίνητοι. Είναι δυσκίνητοι όμως επειδή είναι δημοκρατικοί. Και επειδή είναι χρειάζεται χρόνο. Και εδώ ακριβώς πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή να υπάρχει νομιμότητα η οποία απαιτεί χρόνο αφενός, αλλά αφετέρου να λύνουμε προβλήματα ταχαίως, ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Για το εξάμεινο. Δεν θέλω να σας μπερδέψω με αυτό. Όταν αντιμετωπίζουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα της ασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας, και αν δεν ε, παρερμηνεύω τις φυγουμετρήσεις στο Ευρωβαρόμετρο, ε, για το θέμα αυτό της ασφάλειας έχουμε τους πολίτες με το μέρος μας. Σε κάθε χώρα, από τα 17 και πάνω χρόνια, όλοι θέλουν ε, ένα πιο συντονισμένο μηχανισμό δράσης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ασφάλειας. Αν τα εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουμε δυσκολία να εξασφαλίσουμε αυτές τις αλλαγές που χρειαζόμαστε νομιμοποιούμαστε απόλυτα λόγω των συνθήκων. Ε, στο, εξάμεινο, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο έχουμε αυτή τη διαδικασία της α, ε, αξιολόγησης από ομοτήμους. Βάζεις, ας πούμε, ο καθένας βάζει τα, τα δεδομένα του επιτάπητος ε, και αξιολογείται από τους άλλους. δεν είναι υποχρεωτική αυτή η αξιολόγηση, αλλά πραγματικά υπάρχει η λογική του, της τηλίτευσης για όποιον δεν κάνει τη δουλειά που έχει αναλάβει να κάνει, ας πούμε. Το ίδιο και στην κλιματική... Α, το ίδιο δεν είναι στην, με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό εκεί. Ενώ στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, υπάρχει η αξιολόγηση, η αξιολόγηση από ομοτήμους. Ε, αξιολογείς από τους ομοτήμους σου και αν δεν έχεις κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, αν δεν έχει μάθει το μάθημά σου, αν έχεις διαβάσει ας πούμε, ε, στιγματίζεσαι, στυλιτεύεσαι. Ε, δεν σε τιμωρεί κανένα διανόμου ας πούμε, αλλά ατιμάζεσαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίος τρόπος για να λειτουργούμε. Ε, και το λέω αυτό γιατί ξέρω από επιστήμη, είμαι επιστήμονας και καταλαβαίνω τι λέω. Νομίζω ότι λειτουργεί ήδη αυτή η λογική. Και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λογική πιο πλατιά. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και πρέπει να εφαρμοστεί σε τομείς που υπάρχει καθυστέρηση. Ε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την επιτάχυνση χωρίς να επιβάλλουμε τίποτα από πάνω. Θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς όπου τα πράγματα κινούνται με συμφωνία. Δηλαδή, γίνεται μία ανάλυση για τα, το τι έχει πετύχει με βάση τις δεσμεύσεις που, έχει, που έχεις αναλάβει. Είναι πολύ ωραίος δημοκρατικός τρόπος αυτός. Και μας δίνει και αποτελέσματα, τα οποία είναι πολύ καλύτερα από αυτά που έδωσαν οι παλιές μέθοδοι. Παλιά υποσχόμαστε θα κάνουμε το τάδε, το δίναμε με βάση το σημείο α ή β κτλ. και κανένα δεν ενδιαφέρονταν για ό,τι έκανε τελικά. Αλλά κάποια στιγμή ε, φτάνουμε στο διατάφτα. Φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι θα αναλάβει τον προπολογισμό με τον άλλων χωρών, με το εξάμεινο δηλαδή. Δεν σου είναι δυνατότητα να επιτάσεις ε, και να διατάσει τις άλλες χώρες ε, για ό,τι θα κάνουμε τον προπολογισμό τους. Αλλά υπάρχει αυτός ο μηχανισμός κινήτρων, ας πούμε, ο οποίος είναι πολύ ελκυστικός μηχανισμός. Ε, και το βλέπω να λειτουργεί και στο τομέα της ασφάλειας και άμυνας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό, αυτή την αξιολόγηση, ας πούμε. Κάθε τρία χρόνια θα μπορούσαμε να την κάνουμε, Φερρυπίν. Τέλο πάντων, ό,τι αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός πιο συχνά, να εφαρμόζεται γενικά πιο συχνά σε διάφορους ε, τομείς. Εγώ το, τον ονομάζω αξιολόγηση από μοτίμους, πέστε το αλλιώς. Τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι εκεί το θέμα. Ε, the, Ποιος βάζει φρένο στην υλοποίηση της Λευκής Βίβλου. Είναι μια, ένα συνδυασμό πραγμάτων και αιτίων. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι ιδέες κυκλοφορούν ε, από τη συνήκη της Λισαβόνας και μετά και λίγο πριν. Όμως, με η επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας έγινε λίγο πριν την κρίση. Δεν υπήρξε επαρκές χρονικό διάστημα. Τότε συζητούσαμε τα πάντα, όλα ήταν ανοιχτά με την ίδια ένταση. Και όταν έφτασε η κρίση, τα μυαλά των Ευρωπαίων ηγετών ήταν λιγάκι ας πούμε σκόρπια. Ε, αντί να ασχοληθούν και να επικεντρωθούν στην κρίση. Το λέω αυτό γιατί σήμερα θα πρέπει να δράσουμε διαφορετικά. Και επίσης, στη γειτονία μας χτύπησαν διάφορα καμπανάκια απίστευτα δυνατά. Κοιτάξτε τη γειτονία μας. Σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση με το τοπίο της ίδιας γειτονιάς το 2005-2006. Τη στιγμή που χτύπησε η κρίση, παράλληλα άλλαξε δραματικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά η γειτονία μας. Και σε όρους ασφάλειας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική κρίση με τους πρόσφυγες λόγω του πολέμου στη Συρία. Εάν η Συρία δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση σήμερα, δεν θα είχαμε μία από τις πιο σημαντικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε συλλογικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά με μεγάλη προσοχή. Ναι, νομίζω. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να γίνει με πολύ πιο ενδελεχή και σοβαρό τρόπο. Νομίζω πως πρέπει να γίνει. Γιατί όχι μόνο η οικονομική κρίση μας έπληξε σαν κεραυνό σε εθρία, αλλά και άλλες κρίσεις που έσκασαν παράλληλα με την οικονομική κρίση ήταν και αυτές ευθνίδιες και αναπάντεχες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εκπλήσεται τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, να την πιάνουν τόσο πολύ στον ύπνο οι διάφορες κρίσεις. Νομίζω ότι απάντησα λίγο πολύ όλες τις ερωτήσεις. Όλες τις σημαντικές ερωτήσεις μου απευθύνατε. Αλλά να σας τονίσω ακόμα κάτι. Το έγγραφο που σας παρουσιάζετε που το ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν είναι δική μου πρωτοβουλία, μου ζητήσατε να το παρουσιάσω, δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο δίνει απαντήσεις. Μιλάει για διαδικασίες και θέτει τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, αλλά δεν δίνει αυτές τις απαντήσεις. Εάν ποτέ θελήσετε τη συμβουλή μου, τα σχόλιά μου, τις απόψεις μου, με χαρά να σας τα δώσω. Αλλά σας παρακαλώ, άλλο οι απόψεις μου, άλλο το έργο που σας παρουσιάζω. Μην κάνουμε τη σύγχυση, έτσι, ανάμεσα στα δύο. Ευχαριστώ για αυτή την παθιασμένη παρουσίαση. <laughs> Yes, it was... Ήταν πραγματικά συναρπαστική η παρουσίασή σας και φυσικά δεν φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης για όλα αυτά τα θέματα. Είναι θέματα που θα αποσχολήσουν και το Συμβούλιο στο τέλος του μηνός. Στη συνέχεια θα γίνει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ και βεβαίως όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν. Και να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι πριν από το Συμβούλιο θα διοργανωθεί και το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμείς εκφράζουμε βεβαίως την ελπίδα μας ότι η Μεγάλη Βρετανία θα παραμείνει στην οικογένειά μας και θα συμβάλλει από τη σκοπιά της σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τροφή για σκέψη όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε αλλά δεσμεύομαι ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για την πολύ ζωντανή συζήτηση που είχαμε σήμερα για όλα τα θέματα της εμείς διάταξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τη Γραμματεία της Επιτροπής ΕΝΤΕ για την προετοιμασία των ε, συνεδριάσεών μας και να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για το πολύ δύσκολο έργο τους σήμερα. Κάποιοι ομιλητέ, συμπεριλαμβανομένου και μου, μιλήσαμε αρκετά γρήγορα σήμερα τις παρεμβάσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ.